Uh, let's start. Ελπίζω να έχει ασχοληθεί κάποιο με τα φώτα, γιατί νιώθω σαν να είμαστε σε θεατρική παράσταση. Ε, αν δεν έχετε παρατηρήσει, ε, ε, κρίνουμε χωρί τροποποιήσει την ε, μέση διάταξη. Έχω κάποιε εξαγγελίε, θα γίνουν ε, δύο έκτακτε συνεδριά ΕΜΒΗ ε, στο Στρασβούργο το Μάρτιο. Τη Δευτέρα στις 12 Μαρτίου στις 7 θα ψηφίσουμε για την έκθεση Λαβία για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Την Τετάρτη 14 Μαρτίου από 2 μέχρι 3.30 θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με, τον... με την κυρία Πιενκόσκα για τη... το follow-up που δίνεται στις συστάσεις ε, της Εξεταστικής Επιτροπής ΕΜΕΣ. Δεύτερον, έχετε μέσα στους φακέλου σας ε, τις εκθέσεις ε, αποστολών από τις αντιπροσωπείες στο Πόρτο Μαγκέρα και ε, στην Πάρμα για τον Εύσα. Με τρίτον, μετά την αναπομπή από την Ολομέλεια για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. ο πρώτος τριμερής θα λάβει χώρα αύριο το πρωί με τον εισηγητή Μπά Έικχαρτ, θα είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου για την εισηγητή. Θα πηγαίνει στους τριμερείς και στις παρασκευαστικές συνεδριάσεις για τα θέματα όπου εμείς έχουμε ε, αποκλειστική αρμοδιότητα. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και είναι και διαθέσιμο ε, τα έγγραφα ηλεκτρονικά ως συνήθως ε, αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Κατόπιν. Συστάσεις των συντονιστών ε, σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη συνεδρίασή του 20 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν συστάσεις ε, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Το ίδιο για τα πρακτικά της συνεδρίασής μας 11 Ιανουαρίου. Εάν δεν τυπώσετε ενστάσεις ε, μέχρι το πέρα της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Καλά μου φαίνονται τα πράγματα με τα φώτα, αλλά ακούω περίεργους θορύβους. Για τις ε, προϊόντες ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις να πω ότι ο, ένας δεύτερος και τελευταίος άτυπος τριμερής για την ε, έγκριση και την ε, εποπτεία των ε, φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κοινιατρική κρίση και για την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έγινε στις 21 Φεβρουαρίου. Καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για όλα τα στοιχεία, τα σημεία. Όμως, όπως αποφασίστηκε και στον πρώτο τριμερή, ε, θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία μόλις ε, καταλήξουμε σε έγκριση και για τον ε, φάκελο VMP και μπορούμε να ολοκληρώσουμε δηλαδή την τεχνική ευθυγράμμιση των προτάσεων για τα δύο ζητήματα. Για την πρόταση κα, κανονισμού για την Ενεργειακή Ένωση οι συζητήσεις στον πρώτο άτυπο τριμερή βασίστηκαν στη δική μας θέση, θέση που κρίναμε στις 17 Ιανουαρίου, και τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου της 18 Δεκεμβρίου, επικαιροποιημένη σε σχέση με την πλειοψηφία των δικών μας τροπολογιών. Κάναμε την πρώτη ανταλλαγή, όπως σας είπα, για τα πλέον σημαίνοντα πολιτικά ζητήματα στην πρόταση και ε, παρουσιάσαμε τις ε, συμφωνίες, τα σημεία συμφωνία και διαφορά ε, και στη συνέχεια συζητήσαμε για διάφορε διατάξει σε τεχνικό επίπεδο. κάναμε απογραφή των αερίων θερμοκήπιου, τη προ τις διατάξεις σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων, για την προσαρμογή, για το, την οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη στις αντισόμενες χώρες και ε, διάφορες τροπολογίες για το ETS, για τη, το effort sharing και και ε, τις ε, τροπολογίες σε σχέση με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Ας περάσουμε τώρα στο πρώτο σημείο της σα διάταξη ε, σχέδιο δράσης ε, για την ε, μικροβιακή αντοχή. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την Κάριν Κάντενμπαχ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολλά και στην Επιτροπή μας και αποτελεί και κεντρικό σημείο πολλών ε, δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, δραστηριοτήτων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει πάρα πολλέ συζητήσει. Τα τελευταία χρόνια έχουν ε, συσταθεί διάφορα σχέδια, δράσης. δράση. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό αναφέρεται η έκθεσή μα. One Health φορείται και υπάρχουν διάφορε δράσει, διάφορε οδηγίε που εν μέρη πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη, ε, κυρίως αυτά όπου υπάρχει μεγάλη στέρεση. Ε, θα πρέπει να ε, δούμε και κάποια νούμερα για τη μικροβιακή αντοχή. Τι σημαίνει η μικροβιακή αντοχή λοιπόν σημαίνει ότι τα φάρμακα, τα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν λειτουργούν πλέον για διάφορα μικρόβια. Εάν συνεχίσουμε έτσι, ενδέχεται σε κάποια χρόνια Ε, κάποιες ε, παραδείγματος χάρη λοιμώξεις του αναπνευστικού να, να είναι θανατηφόρες σε λίγα χρόνια ή όταν γίνεται ε, παραδείγματος χάρη Οι μεταμοσχεύσεις επίσης ε, μπορούν να είναι θανατηφόρες λόγω της αντίστασης σε κάποια μικρόβια. μιλάμε επίσης Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο σε 700.000 θανάτους που μπορούν να αποδοθούν σε ε, αυτή την μικροβιακή αντοχή. Ε, κανείς όμως δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους και υποψιαζόμαστε ότι είναι πολύ υψηλότερη η αριθμή. Επίσης υπάρχουν οι λοιμώξεις που σχετίζονται με φαρμακευτικές αγωγές. Είναι κάποιος ας πούμε σε ένα γυροκομείο ή σε ένα νοσοκομείο και ακολουθεί μία ε, φαρμακευτική αγωγή ε, και ένας ιός, όχι ιός, όχι ιός, λάθος το είπε, ε, κάποιο παράσιτο προσβάλλει τον οργανισμό του και τα, η αντιβιωτική αγωγή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. 37.000 θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι υποψιαζόμαστε είναι πολύ υψηλότερα τα νούμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό ε, συνιστά πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τον ασθενή γιατί δεν είναι αποτελεσματική η φαρμακευτική αγωγή, για το σύστημα υγείας συνεπάγεται αυτό πολύ υψηλότερες δαπάνες. Έχει γίνει μια εκτίμηση από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ένα λεπτό γιατί δεν έχω μπροστά μου το νούμερο δυστυχώς για να σας το πω. Μέχρι το 2005 έχει εκτιμηθεί ε, ότι ε, οι δαπάνες θα ανέλθουν ε, στο ίδιο επίπεδο με τις απώλειες που είχαμε με την οικονομική κρίση του 2008 εάν δεν κάνουμε κάτι κατά της μικροβιακής αντοχής. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση της μικροβιαϊκής ε, αντοχής. Από τότε που αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε την πενικυλίνη, θεωρήσαμε ότι βρήκαμε την πανάκια, το ε, τη θαυματουργή ε, φαρμακευτική αγωγή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει υπερσυνταγογράφηση, υπέρχρηση, κατάχρηση των αντιβιωτικών χωρίς να προηγείται μια ξεκάθαρη διάγνωση και ε, βλέπουμε ότι ε, είναι πάρα πολύ σύνηθες ε, Κάποιο ε, που έχει προσβληθεί από έναν ιό να πηγαίνει στο φαρμακείο, να πηγαίνει στον γιατρό και να επιμένει να του συνταγογραφήσει αντιβιωτικό να ασκεί αυτή την πίεση χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί χάρη σε εξετάσεις ότι χρειάζονται αυτά τα αντιβιωτικά και υπάρχει και η... Η αυτοΐαση, ε, ε, η χρήση αντιβιωτικών που, υπάρχουν ήδη, που έχουν ήδη ασθενείς είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα ε, και βλέπουμε ε, ότι και σε εκτινιατρικό επίπεδο υπάρχει κατάχρηση των αντιβιωτικών για, μεγαλύτερη, για πρόληψη και για μεγαλύτερη ανάπτυξη του ζωικού κεφαλίου και αυτό ε, είναι μια τάση που εντείνεται τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πως ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αυτό το γεγονός και στις διαπραγμάτευσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες γιατί ε, η χρήση αντιβιωτικών ε, στην εκτροφή για προληπτικούς λόγους είναι κάτι που θα πρέπει να απαγορευτεί και ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης όλες τις σχετικές συστάσεις. Μέρη τις έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου. Ε, και αναφέρουμε σε αυτό το δεύτερο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα σήμερα ε, με σαφήνεια να πω ότι για μένα τουλάχιστον είναι λείπει το ψαχνό, δηλαδή ε, υπάρχει ένα σκελετός αλλά θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά, να εμβαθύνουμε σε πάρα πολλές ε, προτάσεις γιατί είναι πάρα πολλοί τομεί ο οποίους πρέπει να δράσουμε, χρειάζεται καλύτερη διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής αλλά και σε επίπεδο ασθενών, δηλαδή health literacy, ε, χρειαζόμαστε ξεκάθαρα σχέδια, κριτήρια συγκεκριμένα βάσει των οποίων θα γίνεται η συνταγράφηση ε, όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για κτηνιατρική χρήση ε, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν οι αρνητικές επιπτώσεις ε, το, της ε, και κατάχρησης ε, των αντιβιωτικών στην εκτροφή. Παιδεία λοιπόν, ενημέρωση, πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι τι κάνουμε με αυτά τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά. Μήπως θα μπορούσαμε με κάποιες δράσεις να δούμε ποιες είναι οι ενεργές ουσίες ε, ούτως ώστε ε, αν ξέρουμε κάτι και αν ξέρουμε ότι έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα να παραμείνει στην αγορά και τα υπόλοιπα φάρμακα να αποσυρθούν και χρειαζόμαστε και νέα φάρμακα, νέα αντιβιωτικά ε, που θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα θέλουμε το ελάχιστο δυνατό να χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά φάρμακα, ε, ταυτόχρονα όμως θέλουμε νέα φάρμακα. Καταλαβαίνετε ότι για τις φαρμακευτικές εταιρείες χρειάζονται πολύ ψηλά ποσά για την έρευνα, για να βρουν νέα μόρια, νέα ε, νέες δραστικές ουσίες ε, και ταυτόχρονα θέλουμε να μειωθεί η χρήση των αντιβιωτικών. Βλέπουμε ε, ότι σε αυτό το τομέα και σε άλλους ε, χρειάζεται υποστήριξη για να προωθήσουμε τις θέσεις μας οι οποίες είναι και αμφιλεγόμενες. Ε, θα ήθελα ήδη να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες που μου έχετε στείλει και για τις συστάσεις σας. Α, και κάτι άλλο, ένα τομέας ε, που δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία του είναι η πρόληψη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πολύ καλά προληπτικά μέτρα, εμβολιασμό σε παραδείγματο χάρη, ε, που βοηθά το νοσοποιητικό σύστημα Χρειαζόμαστε παιδεία, διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση, όπως σας έλεγα και σε αυτό το τομέα και ε, σε στενή συνεργασία με τον ε, ΕΜΗ, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, με τον ΕΕΦΣΑ, με το Κέντρο Παρακολούθησης των Λιμωδών Νοσημάτων για να ε, γίνεται η κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη, να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ούτως ώστε να διοχετεύσουμε τους πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς αυτούς τους οργανισμούς για να επιτελέσουν το έργο τους. Νομίζω ότι επί τη βάση αυτού αυτού του σχεδίου που σας καταθέτω θα μπορέσουμε μόνο από κοινού να δράσουμε και από ε, πλευράς ελικοτεχνικής υποστήριξης και από πλευράς σχεδίων δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Μόνο έτσι θα έχουμε τα επιθυμητά αποτέλεσμα και ε, θα πρέπει να αναδειχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα γιατί πέρα από την απειλή για την δημόσια υγεία ε, θα βαρύνει με δραματικό τρόπο τρόπο τα δημόσια οικονομικά τα, επόμενα έτη ε, και θα πρέπει σε όλους τους τομείς ταυτόχρονα να καταλήξουν οι προσπάθειές μας όχι μόνο στο, για τα ανθρώπινα φάρμακα αλλά και για τα ανθρώπινα για ακτινιατρική χρήση ε, και να μην ξεχνάμε ότι Υπάρχουν και αυτές οι νοσοκομιακές ε, λοιμώξεις, όπως είπαμε, ένας ε, ε, τομέας που επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς και η αλυσίδα τροφίμων, που όπου λόγω ενημέρωσης υπάρχουν εξίσου σημαντικά προβλήματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μας έδωσαν δεδομένα από την από τον τομέα της γεωργίας, από τον τομέα της έρευνας, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να επιληθούν ε, το ζητήματο το ταχύτερο δυνατόν ε, να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα ούτω ώστε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο να προωθήσουμε αυτή τη θέση μας όταν διαπραγματευόμαστε εμπορικέ συμφωνίες με τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε κάποια χρονικά όρια διότι έχουμε προσκελέστατο κατάλογο ομιλητών. Όταν βλέπετε τα αστεράκι να βοσβήνει, φαίνεται ότι έχετε περάσει ήδη το χρόνο σας. Ο κύριος Πέτερλε, εκ μέρους της κυρίας Ζόμερ. Ευχαριστώ. Τιμή και προνόμιο για μένα να είμαι σαν Αλόης Ζόμερ, σαν εισηγητής του σκιώδους εισηγητού. Θα έρθει αργότερα όμως. Θέλω να παρουσιάσω αυτά που ετοίμασε η σκιώδη συγγήτρια, η κυρία Ζόμερ. Είναι πολύ ικανοποιημένη από την ισορροπημένη ε, έκθεση της κυρίας Κάλεμπαχ. Την ευχαριστώ γι' αυτό. Η συγγήτρια αναφέρθηκε στα σημαντικότερα θέματα. Πιστεύει ότι κατεπηγόντως χρειαζόμαστε νέα αντιβιωτικά. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να αναπτυχθούν νέα αντιβιωτικά. Η παραγωγή είναι μακροχρόνια και πολύ δαπανηρή χρειάζεται περίπου 20 χρόνια ανάπτυξη νέου αντιβιωτικού. Το μεταξύ αναπτύσσονται νέε αντιστάσει. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για την παραγωγή νέων αντιβιωτικών. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειαζόμαστε υπεύθυνη χρήση των υφισταμένων αντιβιωτικών. Τα αντιβιωτικά συχνά λαμβάνονται σε υπερβολικέ ή με εσφαλμένο τρόπο. 30-50% των συνταγωγημένων αντιβιωτικών περιτεύουν και πολύ γρήγορα τα χορηγούν οι γιατροί. Πολύ συχνά οι ασθενείς ε, παίρνουν με λαθασμένο τρόπο αντιβιωτικά ή τα σταματάνε πολύ νωρί. Δεν είναι καλά ενημερωμένοι περί αντιβιωτικών οι Ευρωπαίοι. 57% αυτών δεν γνωρίζουν ότι δεν επηρεάζουν καθόλου ε, τους ιούς τα αντιβιωτικά. Και ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιωτικό πυρετό ε, που παράγεται από έναν ιό. Και θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόληψη. Η αύξηση της αντιμικροβιακής αυτής αντίστασης προέρχεται στην ε, κακή υγιεινή στο σύστημα ε, υγείας, κυρίως για βάλλοντε ομάδες. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την πρόληψη των μολύνσεων. Χρειάζεται μέσω εμβολιασμών ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα και είναι αποτελεσματικό πλευρά κόστου. Είναι υποφελέ οικονομικά. Επίση, τεράστια χρήση αντιβιωτικών στα ζώα στι εκμεταλλεύσει παίζει σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται σωστή στέγαση των ζώων και κτηνιατρική μέρημνα και ισορροπημένη διατροφή. Όλα αυτά μπορεί να συμβάλλουν στην υγεία των ζώων και να μειωθεί η χρήση των αντιβιωτικών. Θα πρέπει να υπάρξουν και εναλλακτικέ λύσει αντί των αντιβιωτικών. Η αντιμικροβιακή αντίσταση είναι πραγματικό πρόβλημα κοινωνικό και οικονομικό. Κάθε χρόνο 25.000 άνθρωποι στην Ευρώπη και 700.000 άνθρωποι στον κόσμο πεθαίνουν από αυτή την αντιμικροβιακή αντίσταση. Σύμφωνα εκτιμήσει, θα αυξηθούν κατά πολύ αριθμοί τα επόμενα έτη. Μπορεί να έχουμε 10 εκατομμύρια θανάτους από αυτό το αίτιο το 2050, πάνω από αυτούς που πεθαίνουν τώρα από τον καρκίνο. Είναι η ώρα της δράσης. Προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια και τους σκιώδης. Και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπιέκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία, εισηγήτρια, Κυρία Συγήτρια, παρουσιάσατε το σχέδιο εκθέσεώς σας λεπτομερέστατα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσεως για την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντιστάσεως είναι ε, κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί κατεπήγον. Η, η μη ορθή χρήση των αντιβιωτικών, η υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών και κακός έλεγχος στον τομέα των αντιβιωτικών, όλα αυτά οδηγούν στη σημερινή κατάσταση που είναι πολύ επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την υπερβολική χρήση ελαφρά την καρδία των αντιβιωτικών, διότι μέσω αυτής της υπερβολικής χρήσεως η αποτελεσματικότητα των αντιβιωτικών μειούται και ε, αναπτύσσονται νέα μικρόβια τα οποία ε, έχουν μεγάλη αντίσταση στα φάρμακα. Προφανώς πρόκειται περί αντιβιωτικών επίσης που χρησιμοποιείται και στα ζώα. Ισχύει αυτό. Πέρα από την ε, δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα παγκόσμιο θεματολόγιο κατά πολεμήσεως της μικροβιακής ε, αντίστασης. Σήμερα υπάρχουν σχέσεις στενές μεταξύ των χωρών. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε απομόνωση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάντα τα μικρόβια διέρχονται τα σύνορα. Χρειάζεται λοιπόν μια διεθνή συνεργασία. Θα έπρεπε επίσης και η ευρωπαϊκή δράση να λαμβάνει υπόψη τον κατάλογο με προτεραιότητες που έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσον αφορά τις παθογόνες ουσίες. Και θα πρέπει να αποφύγουμε την επιστροφή κάποιων ασθενειών όπως είναι η φυματίωση παραδείγματος χάρη και κάποιες δυσμονισμένες ασθένειες που επανακάμπτουν σήμερα. Έχω την εντύπωση έχουμε την εντύπωση ότι λύσαμε μέσω εμβολίων προβλήματα, αλλά επανέρχονται παλιέ ασθένειες και πάλι. Εκτιμούμε ότι μέχρι 100 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν λόγω της αντίσταση ε, αντίστασης ε, στα αντιβιωτικά από τώρα μέχρι το 2050. Και προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα απώλειες που θα αντιστοιχούν στις οικονομικές απώλειες της κρίσης του 2008, της οικονομικής κρίσης παγκόσμιας του 2008. Πάμε κάνουμε τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ναι, μιλάω εξ ονόματος της Λίντα Μπόιλε και θα ήθελα να πω ότι ε, όλα αυτά είναι, οι στατιστικές δηλαδή που έχουμε ακούσει είναι πραγματικά ε, ε, εκφοβιστικές για κάποιον που μπαίνει ξαφνικά μέσα στην αίθουσα. Βεβαίως υπάρχει σχετική δράση αλλά μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να υποστηριχθούν περισσότερο και οι δράσει στα κράτη-μέλη. Ε, ζητούμε δράση έτσι ώστε να υπάρχει ένα σωστό ε, σχέδιο δράσης ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μικροβιακή αντοχή. Ε, ένα σχέδιο δράση λοιπόν, επί των οποίων εγώ θα υποβάλω κάποια σχόλια μέσω τροπολογιών. Πρώτα απ' όλα ε, ασχολούμαστε με περιβαλλοντικά θέματα και δημόσια υγεία. Γι' αυτό λοιπόν είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι υπάρχει τόσο λίγη δράση όσον αφορά το περιβάλλον. Ε, το πρωτόκολλο το οποίο σχετίζεται με το θέμα αυτό προβλέπει συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ε, υποβάλει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα στην έκθεση αυτή. Δεύτερον, όσον αφορά τους σπόρους, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συγκεκριμένη στοχοθέτηση από πλευράς των κρατών μελών με υπολογισμό του κόστους. Η παρούσα κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Προσπαθούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τη μικροβιακή αντοχή με ίδιους σπόρους και ο καθένας με τον τρόπο από το Εμείς θέλουμε ενοποιημένα πρότυπα και ε, αποδοχή ε, πόρων όσον αφορά ε, το θέμα αυτό τελικό μου θέμα σχετίζεται με την ανάπτυξη της έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ευρωπαϊ... έχει ηγετική θέση όσον αφορά ε, την ε, έρευνα κατά της μικροβιακής ε, αντοχής. Ο... Δεν είναι δυνατόν όμως να προχωρήσουμε την... στην κατάσταση αυτή όπου δεν γίνεται καινούργια έρευνα όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Και ούτως ή άλλως αυτό το πρόβλημα θα εμφανίζεται μπροστά μας διαρκώς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό της ε, ε, μικροβιακής ε, αντοχής μέσα από ανάπτυξη νέων σύγχρονων και καινοτόμων τρόπων γρήγορης διάγνωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. To see if uh, the other shadows are here. Να δω, λέει η Πρόεδρος, Ε, αν είναι εδώ ε, άλλοι σκιώδεις, είστε σκιώδεις. Α, δεν σας είδα, ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαι ακριβώς ε, ε σκιώδης, αλλά προσωπώ τον συνάδελφο ο οποίος καθυστέρησε λίγο. Θα μιλήσω στα Σουηδικά, γιατί θα πω τις απόψεις του και και θα ήθελα να μεταφέρω τις απόψεις του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο δράσης εντόπισε τις μεγαλύτερες ε, προτεραιότητες ε, της καταπολέμησης ε, αυτού του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής. Όμως δεν καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Πώς πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό εμείς ε, θα πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ζητάμε ε, μεγαλύτερη πυγμή και περισσότερες ε, προτάσεις. Αυτά σε γενικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα σε όλους τους τομείς Ε, και μην ξεχνάμε το 70% της ε, μικροβιακής αντίστασης οφείλεται σε κτηνιατρική χρήση φαρμάκων. Επίσης, ε, η διάδοση αυτών των ανθεκτικών μικροβίων οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις νοσοκομιακές λοιμώξεις και στην κακή υγιεινή. Ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρειαζόμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένα μέτρα. Όμως, ε, δεν φτάνουν τα νομοθετικά μέτρα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή Υπάρχουν, παραδείγματο χάρη, κριτήρια ε, που σχετίζονται με την καταπολέμηση μικροβιακή ε, αντοχή ε, όταν σερβίρεται, παραδείγματο χάρη, κρέα στα νοσοκομεία ή στα σχολεία. Θα πρέπει επίσης να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναδείξει σε προτεραιότητα αυτό το θέμα στις ε, διαπραγματεύσεις ε, διεθνών συμφωνιών. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, συνάδελφο, ε, για την εργασία της. Οπωσδήποτε η κατάσταση είναι κατεπίγουσα αυτό της μικροβιακής αντοχής. Αλλά ε, ε, στα πλαίσια της αρχής της μίας υγείας επί της οποίας βασίζεται η έκθεση πιστεύω ότι όσον αφορά την στρατηγική για την κτηνοτροφία δεν έχουμε αναπτύξει τόσο καλά το θέμα. Στην παράγραφο 2 γίνεται λόγο στην κτηνοτροφία και την κτηνοκαλλιέργεια. Ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούν τα όσα υπόθηκαν ε, κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων ε, για την δικιά μου έκθεση για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Στην παράγραφο 11 ε, γίνεται λόγος για την, για την απαγόρευση πώλησης αντιβιωτικών φαρμάκων από τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο, ο, από, συγγνώμη, από τους κτηνιάτρους. Ωστόσο, οι κτηνίατροι σε πολλές περιπτώσεις είναι οι μοναδικοί που μπορούν να παράσχουν τα φάρμακα αυτά όταν σε ακτίνα μέτρων δεν υπάρχουν φαρμακεία. Επίσης, ε, ε, κινητροδότηση για την έρευνα. Ε, κίνητρα για την έρευνα όπως κάναμε και για τα ορφανά φάρμακα και για τα παιδιατρικά φάρμακα. Είμαι απολύτως υπέρ των παραγράφων 9 και 10 που υπογραμμίζουν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα εργαλεία έγκαιρης διάγνωσης για τα μικροβιακά στελέχη και την αναγνώρισή τους και τέλος στις παραγράφους 27 και 28 επιμένουμε στην ανάγκη παρέμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να επιβάλλουμε την αμοιβαιότητα των προτύπων μα όσον αφορά ε, τι ε, εισαγωγέ κτηνιατρικών ε, διορθώνω κτηνοτροφικών εισαγωγών και επίσης να απαγορεύσουμε σε, στα σφαγεία να χρησιμοποιούν οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια απαγορεύονται ή στην Ευρώπη. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ. Ναι, είναι γεγονός ότι χρειάζεται αμοιβαιότητα όσον αφορά τα τρόφιμα ε, τα οποία εισάγουμε στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση ε, στην ε, έκθεση της Κομισιόν εκεί που λέει ότι απειλούνται οι πρόοδοι λόγω της καταχρηστικής ή ε, ε, μη δέουσας χρήσης των αντιβιωτικών που έχουν οδηγήσει στην χρήση, ε, στη γνώμη, στην εμφάνιση και τον πολλαπλασιασμό ανθεκτικών στα αντιβιωτικά στελεχών. Αυτό τι σημαίνει και εδώ μπορώ να συμφωνήσω με την εισηγήτρια την οποία θα ήθελα λοιπόν, να συγχαρώ για την έκθεσή της. Χρειάζεται επομένως πρόληψη, μια πολιτική πρόληψη στη Γαλλία. Είχαμε ξεκινήσει μια εκστρατεία για τα αντιβιωτικά όταν πρέπει και μόνο όπως πρέπει. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπαιδεύσουμε και τους ασθενείς και τους πολίτες οι οποίοι πάντα ζητούν τα αντιβιωτικά λες και είναι πανάκια και θαυματουργό φάρμακο για όλα. Θα πρέπει να ασκηθεί η πίεση λέμε και για τους ε, ε, ασθενείς ανθρώπους αλλά και για την κτηνοτροφία. Ε, εγώ θα ήθελα και το θέμα αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως των κτηνιατρικών φαρμάκων να οδηγηθεί κάπου γιατί εκεί συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με την έλογη χρήση των κτηνιατρικών αυτών φαρμάκων. Επίσης, όσο πιο πολλές εντατικέ κτηνοτροφικέ μονάδες αναπτύξει κανείς, τόσο πιο πολύ θα πρέπει να δράσει στο προληπτικό σκέλο. γιατί εκεί θα, παίξουν, θα παίξει μεγάλη σημασία το θέμα της μη διάδοση των ασθενών, ασθενειών. Από άποψη ε, οικονομική θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα στοιχεία, όχι μόνο το κόστος των ε, αντιβιωτικών, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και εναλλακτικέ λύσεις, φαγοθεραπεία ας πούμε, η οποία είναι συμπληρωματική της ε, χρήσης των αντιβιωτικών. Έχετε ας πούμε έναν ε, κιανού και σε αυτή την περίπτωση έχει αναπτυχθεί ισχυρή αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, φάρμακα τα οποία μπορούν, ε, στην Ευρώπη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ε, γεωργία α πούμε και επομένως στην ουσία δημιουργείται μια, ένα συγκεκριμένο κοκτέιλ ιών που θα δράσει πάνω σε, μια, σε ένα συγκεκριμένο βακτήριο. Ε, βεβαίως μπορεί κανεί να διευρύνει το φάσμα των αντιβιωτικών αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν και άλλε εναλλακτικέ δυνατότητε. Όπω αυτή τη φαγοθεραπεία. Ε, έχουμε ξεκινήσει στην Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά εξαρτώμεθα υπερβολικά από τρίτε χώρε και χώρε οι οποίε δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχά την κυρία Κάλενμπαχ για το σχέδιο εκθέσεώς τη. Αναφέρθηκε σε δύο βασικά σημεία, κυρία Κάλενμπαχ και θέλω να τα αναλύσω περαιτέρω. Και θέλω να δούμε την περιβαλλοντική και την γεωργική πτυχή. Όσον αφορά την αντιμικροβιακή αντοχή, πολλέ φυλάμε για τη χρήση τη χρήση αντιβιωτικών σε ανθρώπινη κλίμακα, αλλά χρησιμοποιούνται και στα ζώα. Και αυτό επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, επηρεάζει και το περιβάλλον. Και αυτό με ανησυχεί πολύ. Αν ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση στον κόσμο το 2015, σε αντίστοιχη έκθεση, λέει δύο τρίτα των αντιβιωτικών που παράγονται σε παγκόσμια κλίμακα κάθε χρόνο, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα στα ζώα. Γνωρίζουμε επίσης ότι όταν τα ζώα καταναλώνουν αντιβιωτικά, 30 με 90% από τα αντιβιωτικά απευθυνόνται μέσω της κοπριάς και των ούρων. Και αυτό μολύνει το περιβάλλον με αντιβιωτικά και με βακτηρίδια τα οποία έχουν αναπτύξει μικροβιακή αντοχή και τα ζώα καταναλώνουν αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά μπαίνουν και στο κρέας και στο γάλα τους. Όλα αυτά καταναλώνονται από τον καθένα από εμά, ακόμα και από τα παιδιά μας. Όταν μιλάει κανείς στου εκλογεί και στους πολίτε τη χώρα μας, βλέπετε ότι ευαισθητοποιούνται για το θέμα και ανησυχούν μάλιστα για την αύξηση τη ε, μικροβιακής αντοχής. Και θα πιέσουν τους λαμβάνοντες αποφάσεις και τους καλλιεργητές και θέλουν τα προϊόντα να προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παίρνουν αντιβιωτικά. Και αυτή η πίεση συνεχώς θα αυξάνεται για κάτι τέτοιο. Βλέπω αυτή την έκθεση λοιπόν. Την θεωρώ θετικά, με θετικό όμα, διότι νομίζω ότι θα καλύψει άλλα θέματα. Δηλαδή πώς να προστατευτούμε και εμείς και τα παιδιά μας. Πώς να εξασφαλίσουμε ότι στο τραπέζι μας βάζουμε ασφαλή φαγητά. Και εφόσον είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να απευθύνω ερώτημα άμεσα προ την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ σχεδιάζει να βοηθήσει του πολίτε πάνω σε αυτό, τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Τέλο, για το περιβάλλον. Όλοι μας θα θέλαμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει με την απελευθέρωση και διάθωση των οργανισμών με μικροβιακή αντοχή στο περιβάλλον. Και μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ερευνήσει τι γίνεται στη σχέση μεταξύ υγεία των ζώων, τι, γίνεται, τι πρακτικές ακολουθούνται στις εκμεταλλεύσεις και πώς αυτά σχετίζονται με τη μικροβιακή αντοχή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιούλερ θα έχει το λόγο. Κυρία Κάντεμπαχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν διεξοδικότατη και εξισορροπημένη η θέση σας στο σχέδιο που μας καταθέσατε. Καλωσορίζω τη θέση σας ε, και χαίρο που, χαίρομαι που δεν κατονομάζουμε εδώ ε, υπευθύνου ε, και υπόπτους, αλλά προσεγγίσουμε με, με ρεαλιστικό τρόπο τα προβλήματα και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε λύσεις έχοντας εντοπίσει τα προβλήματα. Ε, βλέπουμε ε, τι γίνεται στην ανθρώπινη ιατρική, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό, γιατί στην εκτροφή ζωικού κεφαλαίου και στην κτηριατρική χρήση φαρμάκων παρατηρούνται πολλά προβλήματα. Βλέπουμε ότι Υπάρχουν και προβλήματα όπως ε, διάθεση φαρμάκων στα υπόγεια ύδατα ε, και ε, θα ήθελα να ξέρω τι θα γίνει με τον καθαρισμό λιμάτων, δηλαδή ε, στα, στη, στη, στα νοσοκομεία δεν ε, απαιτείται αυξημένο επίπεδο καθαρισμού και βλέπουμε ότι το σύστημα διοχέτευσης των λιμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ούτως ώστε ε, να υπόλοιπα κατάλοιπα αυτών των φαρμάκων κυρίως προέρχονται από νοσοκομεία να κατευθύνονται απευθείας σε σταθμούς καθαρισμού λιμάτων. Ε, πολλά μπορούμε να κάνουμε επίσης και στον τομέα της πρόληψης. Ε, υπάρχει και ένα θέμα που θα ήθελα να τονίσω όλους ιδιαίτερως. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση ανάμεσα στα ζώα εκτροφής και τα οικόσιτα ζώα και θα ήθελα, ε, κατά κατοικίδια δηλαδή ζώα και θα ήθελα να, στην παράγραφο 12 να διευκρινιστεί αυτό. Όταν μιλάμε για τη χορήγηση φαρμάκων από τους κτηνιάτρους θα πρέπει να προβάλλω ένσταση, διότι σε μένα, εγώ είμαι στην Ήπεθρο, 40 χιλιόμετρα μακριά είναι ο κτηνίατρος. Όταν αρρωστήσει η αγελάδα μου, τι θα κάνω, θα πρέπει να ε, οδηγήσω 30 χιλιόμετρα για να ε, πάω να βρω τον κτηνίατρο και να πάω μετά στο φαρμακείο και ε, πώς θα χορηγηθεί το φάρμακο. Δηλαδή δεν γίνεται στην πράξη αυτό γιατί από υψηλό πυρετό θα πεθάνουν όλα τα ζώα πριν προλάβουμε εμείς να φέρουμε τα κατάλληλα φάρμακα. Θα ήθελα λοιπόν από αυτή την άποψη να καταθέσω τροπολογίες και είναι η μόνη αντίρρηση που έχω. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Στρέικ Πέρικ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ε, Κάντενμπαχ. Αυτό το θέμα ε, ε το, μας απασχολεί στις κάτω χώρες εδώ και χρόνια. Ε, επιστημονικές έρευνες ε, έχουν ε, δείξει ότι η μεταβίβαση μικροβίων από το ζώο στον άνθρωπο και η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής είναι πηγές σοβαρών προβλημάτων. Αυτό αντιμετωπίζεται, εντοπίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχουν γίνει και κάποια βήματα. Ε, στον κτηνιατρικό ε, τομέα έχει μειωθεί κατά 65% η χρήση των φαρμάκων. Για τα κατοικίδια ζώα χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο, ε, πολύ ευρύτερα τα αντιβιωτικά από ότι για τους ανθρώπους. ο άνθρωπος παραμένει, ε, συγγνώμη, ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι πλέον ο βασικός μικροβιοφορέας. Ε, τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι ακριβή, είναι πολύ υψηλότερα τα πραγματικά στοιχεία. Είναι ένα ενδυνάμει τσουνάμι ε, τα προβλήματα που οφείλονται στην μικροβιακή αντοχή. Θα πρέπει ε, και στα σπίτια μας αλλά και στα νοσοκομεία να δραστηριοποιηθούμε, να κάνουμε καμπάνιες ενημερωτικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κυρία Κάτενμπαχ, ε, αναρωτηθήκατε ε, πόσο, καιρό θα, πόσο καιρό θα χρειαστεί προτού μια μικρή λίμωξη του αναπνευστικού του ερωποιητικού καταστήθων αντιφόρων. Νομίζω ότι αυτό θα επέλθει πολύ ε, συντομότερα από ό,τι προβλέψατε. Ε, ε, κυρία Γκροστέτ, όπως είπατε, θα πρέπει άμεσα να δράσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Πολύ καλό το κείμενό της, πολύ καλή έκθεσή της πράγματι αντιμετωπίζει αυτό το θέμα της μικροβιακής αντοχής και την προσέγγιση στον τομέα της υγείας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός το κτηνιατρικό ε, τομέα, σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία. Αυτή είναι πολύ σωστή η ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί η έκθεση. Τα επόμενα χρόνια θα συζητήσουμε και άλλη μια πτυχή της μικροβιακής αντοχής. Αυτό που βλέπουμε σε διάφορα κράτη-μέλη όπως είναι η Δανία, αλλά και στην Ολλανδία, και αλλού είναι αύξηση αριθμού εκείνων που μολύνονται από μύκητες από διάφορα ε, βακτηρίδια μύκητες που είναι δύσκολο να θεραπευτούν. Συμβαίνει αυτό στην Ολλανδία και είδα και άλλες περιπτώσεις στη Δανία πρόσφατα. Κινούμεθα προς ελάθος κατεύθυνση λόγω της ε, χρήσεως ε, αντιμικητικών ε, θεραπείων και έτσι είναι πιο δύσκολο να θεραπεύονται οι ασθενείς από μήκητες. Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε και από αυτού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφήνοντας παράμερα αυτό που συζητούμε και αυτό που σα ανέφερα τώρα θα είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο θα έπρεπε να αναφέρετε στην έκθεση. Πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει το ότι θα έχουμε τη δυνατότητα. Αν δούμε ότι ένα προϊόν χρησιμοποιείται ευρύτατα στη γεωργία και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες, τότε αυτό να μπορεί να αποσύρεται, να αποσύρεται η αδειοδότηση, μπορεί να είναι αντιμικητικό, μπορεί να είναι κάποιο αντιβιωτικό, ένα είδος πενικυλίνης. Πρέπει να υπάρχει μια ταχεία διαδικασία που να αφαιρεί ένα πρωί από την αγορά αν χρησιμοποιείται υπερβολικά και αν υπάρχει πόνοι ότι η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν η συγγήτρια να είναι ανοιχτή στο να δώσουμε και κάποιε άλλε πληροφορίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και ο Σπόρτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συγχαίρω την κυρία Κάλεμπαχ, πληρέστατη η προσέγγιση τη. Είμαι βιολόγο και να αναφέρω κάτι που είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Η ανάπτυξη της αντιστάσεως στα αντιβιωτικά είναι φυσική και αναπόφευκτη. Το θέμα είναι ότι επιταχύνουμε τη διαδικασία εμείς. Και αυτό λόγω της συμπεριφοράς μας, της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το χειρότερο που μπορεί να κάνεις είναι να δίνεις μακροχρόνια μικρές δόσεις αντιβιωτικών. Διότι αυτό οδηγεί, διότι οδηγεί σε ανάπτυξη της αντίστασης των μικροβίων. Λοιπόν, προληπτική χρήση των αντιβιωτικών, λάθος. Δεύτερον, η προσθήκη αντιβιωτικών στι ζωοτροφέ. Λάθο. Τρίτον, που αμελούμε η χρήση αντιβιωτικών σαν παρασιτοκτόνο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και η γλυφοσάτη είχε πάρει την άδεια σαν αντιβιωτικό, είχε πατέντα σαν αντιβιωτικό. Πρώτη στη δράση της γλυφοσάτης είναι αντιβιωτική. Πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Η συμπεριφορά μας έναντι φυσικής διαδικασίας φταίει. Επιταχύνουμε τη διαδικασία από τη συμπεριφορά μας. Από εμά εξαρτάται το τι θα συμβεί όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Ο κύριος Πέτερλε. Thank you Σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Νομίζω ότι εδώ έχουμε αρχίσει να σκάβουμε σε ένα ε, παγόβουνο. Και νομίζω ότι η συγγήτρια ακολουθεί τον δρόμο της αληθείας. Και βλέπω ότι η χρήση των αντιβιωτικών πλέον έχει γίνει λαϊκή ιατρική Έχουμε ανθρώπους που μέσω της αυτοίασης δεν χρειάζονται καν γιατρούς ε, και έχουν συνέχεια ε, την ανάγκη για αντιβιωτικά και λένε, αυτή είναι η λαϊκή, το λαϊκό αφήγημα, ότι ο καλός γιατρός γράφει, συνταγογραφεί αντιβιωτικά ε, και τώρα ακόμα και που έχουν γίνει γνωστά όλα αυτά τα στοιχεία ακόμα οι ασθενείς θέλουν διαρκώς να τους γράφει ο γιατρός αντιβιωτικά. Πρέπει να κινηθούμε σε πολλά μέτωπα ταυτοχρόνως. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης νέων αντιβιωτικών. Ωστόσο αυτό που είναι πρώτη τη σημασία κατά την άποψή μου είναι να αλλάξει η, η αντιμετώπιση που έχουμε για τα αντιβιωτικά. Πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις ε, μέχρι τώρα δεν είναι συνολικές ε, και πρέπει να γίνουν ε, και γνωρίζουμε ήδη αρκετά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πριν δημιουργηθούν και σχεδιαστούν νέα αντιβιωτικά ε, και μάλιστα μπορούμε αποτελεσματικά ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα μέσω της ε, των συστημάτων υγιεινής και των συστημάτων υγείας. Ε, η ομάδα εργασίας ε, για την υγεία έχει οργανώσει πρόσφατα ε, κάποια εργαστήρια ακριβώς για το θέμα της μικροβιακής αντοχής, αντοχής δηλαδή κατά των μικροβιοπτών φαρμάκων και το, το πόρισμα λέει ότι μπορούν να μειωθούν οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις μέχρι 70% αλλά ακόμα η κοινή αγορά ή η ενιαία αγορά δεν έχει αγγίξει καθόλου αυτό το κομμάτι της ε, αγοράς. Δεν ασχολείται με αυτά τα προϊόντα, ε, ενώ υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από τα αντιβιωτικά. Ε, θα ήθελα εγώ μια κοινή αγορά η οποία θα λειτουργήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Η κυρία Καμπεδόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Στάνφο Κάρεμπαχ γιατί είναι εξαιρετική η εργασία της. Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα σύνθετο και περίπλοκο, αλλά νομίζω ότι η συγγήτρια κατάφερε μέσα στην έκθεσή της να υπογραμμίσει τα κεντρικά χαρακτηριστικά ε, τα οποία θα μας οδηγήσουν να ε, αντισταθούμε σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας και μάλιστα και να το ξεπεράσουμε. Ε, είναι μια μεγάλη πρόκληση μαζί με την άλλη μεγάλη πρόκληση για την καταπολέμηση του καρκίνου. Πολύ σωστά η συγγήτρια αναφέρεται στις παρούσες ε, ε, ανάγκες είναι σαφές ότι σε τριμερή διάλογο ε, είμαστε πλέον για τα κτηνιατρικά φάρμακα και από εκεί θα πρέπει να προκύψει και ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά την μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών στα φάρμακα και των αυξητικών ορμονών φυσικά κτλ. και γενικώ για, τα, για, τα, για τις φαρμακούχες ζωοτροφές όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, από κοινού. Όσον αφορά ε, την ισορροπία ανάμεσα στη χρήση και την έρευνα, είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε νέας μορφής και γενεάς αντιβιωτικά, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η κακή χρήση, η ελλειπής ή η υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών. Επομένως αυτό το μέτρο θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματική και όσον αφορά την υγεία και όσον αφορά την οικονομία. Πιστεύω ότι η ανάγκη για έλογη χρήση ε, σωστά υπογραμμίζεται στην έκθεση. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο κινήτρων. Ε, τα υφιστάμενα κίνητρα προφανώς ε, δεν είναι τα κατάλληλα όσον αφορά τα αντιβιωτικά και εκεί ακριβώς καταλήγουν όλες οι έρευνες και μελέτες και η μελέτη της Κομισιόν όπου προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία νέων μοντέλων. Η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα πρέπει μέσα από κοινέ και ε, ταυτόχρονες δράσεις να αντιμετωπιστεί. Και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να βασιστούμε ε, και στην τεχνολογία αλλά και στην συνεργασία. Θα πρέπει να υπάρχει και υπερεθνικός οργανισμός ο οποίος ε, θα ελέγχει τα θέματα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει και τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν γιατί είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και πολύ σωστή. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριος Γκέικε. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που συμπεριλαμβάνεται αυτό το θέμα της μικροβιακής αντοχής ε, στο σχέδιο έκθεσής και σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, εμείς εδώ να αποφύγουμε την περαιτέρω ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής και να ασχοληθούμε με το θέμα της έρευνας για τα νέα αντιβιωτικά. Ε, κάτι άλλο που προκύπτει από την τυπώσια συζήτηση στην ε, Γερμανία είναι ε, το περιβαλλοντικό ζήτημα στο, στη Δρέσδη στο Πανεπιστήμιο έγινε μια μελέτη και διαπιστώθηκε ότι στη, στο Σάξεν στα υπόγεια ύδατα υπάρχει μεγάλη μόλυνση από τέτοιους, τέτοια μικρόβια και Καταλαβαίνετε ότι αυτό έσπηρε τον τρόμο στους ανθρώπους και το πιστεύω ότι όπου και να ε, υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα της, ε, ο ίδιος πανικός θα επικρατούσε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφαλείας στην τα Ινστιτούτα επεξεργασία, τα κέντρα μάλλον επεξεργασία ελλημάτων. Χρειαζόμαστε ειδικά φίλτρα με ενεργό άνθρακα, χρειαζόμαστε ε, αντίστοιχη πολιτική στα νοσοκομεία. Αυτά δισεκατομμύρια θα κοστίσουν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο ε, του ε, Δήμου ε, και τι κοινότητε και θα πρέπει με κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συγχρηματοδοτήσουμε αυτέ τι δράσει γιατί τελικά μόνο με τι πράξει επιτυγχάνουμε κάτι και όχι με τα όμορφα λόγια. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται έτσι ο κατάλογος των ομιλητών από τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Τιερή Βενά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρακολούθησα με προσοχή τη σημερινή συζήτηση και εκφράζω την ικανοποίησή μου ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μεγάλο ενδιαφέρον που ε, έχει προκαλέσει το θέμα αυτό γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η δέσμευση τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν ε, ε, υιοθέτησε πέρσι ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης που προέβλεπε και κάποιες δραστηριότητες τις οποίες προτίθεται να αναλάβει. Και για να απαντήσω μάλιστα στην κυρία Νταλή, η οποία μας απίθυνε σχετικό ερώτημα, αυτό το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής ε, αντιμετώπισης και προσέγγισης όσον αφορά τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ε, η παρουσία φαρμακευτικών προϊόντων για το περιβάλλον. Έχει ξεκινήσει ήδη μια σχετική μελέτη η οποία περιλαμβάνει ε, διαβουλεύσεις ε, με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και στόχος πρόθεσή μας είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Πέραν τούτου, για μία ακόμα φορά να πούμε ότι η Κομισιόν ε, εκτιμά σε τη δράση του Κοινοβουλίου και βεβαίως θα μελετήσει προσεκτικά το έγγραφο το οποίο θα παραχθεί από τούτη την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάτεμπαχ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους συνσηγητές, τους σκιώδεις και αυτούς που τους εκπροσωπούν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μας και με όλες τις προσθήκες που έγιναν σήμερα και υποθέτω ότι θα καταθέσετε και συγκεκριμένες τροπολογίες και προτάσεις προσθήκων ε, για το, το σχέδιο. Είμαι πεπισμένη λοιπόν με όλα αυτά θα συμβάλλουμε ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και επίσης θα μπορέσουμε σε επίπεδο κρατών μελών να αποτρέψουμε αυτό το φρικιαστικό σενάριο που αναφέραμε ε, γιατί πέρα από τις συγκρίσεις που κάνουμε με τον καρκίνο και τον αριθμό θανάτων μην ξεχνάμε ότι είναι σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας και σοβαρότατο βάρος για τις οικονομίες των κρατών μελών ε, ε, τα μέτρα σε πολλούς τομείς θα πρέπει να είναι δεσμευτικά. Ένιωσα ότι υπάρχει μια μικρή αντίσταση από τους συναδέλφους, αλλά χρειαζόμαστε νομοθετικά μέτρα και χρειαζόμαστε σωστή εφαρμογή ε, και όχι μονομερή δράση από πλευρά των κρατών μας. ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Η 5η Μαρτίου είναι στι 11 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών και στις 16 και 17 Μαΐου στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε. Για πάμε τώρα στο επόμενο σημείο το eco-design, οικολογικός ε, σχεδιασμός. Ε, η υπηρεσία τεκμηρίως EPRS θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της ε, για την παρακολούθηση εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό. Η συγγήτρια της έκθεσης του Κοινοβουλίου είναι η κυρία Ντομνίκ Φρεντερίκ, συγγνώμη, Πρώτα όμως... Θα δώσουμε το λόγο στο, στην υπηρεσία τεκμηρίωση για την παρα... παρουσίαση της έκθεσης. Η κυρία Ελεονόρ Ντράμπικ, βλέπω, από το CPS θα πάρει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρουσιάσω το έγγραφό μας, το ενημερωτικό τιμάσαμε το φθινόπωρο για το πώς βλέπουμε την οδηγία εμείς διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και ήταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αξιολογήσεως. Επόμενη διαφάνεια. Η μελέτη κάνει μια επισκόπηση της εφαρμογής της οδηγίας. Συλλέξαμε τις απόψεις διαφόρων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι τα θετικά, τα αρνητικά στοιχεία και προβλήματα εφαρμογής. Είχαμε περιγνώμηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κυβερνήσει, κυβερνητικού φορεί 7 κρατών μελών. Εκπροσώπους Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Πορτογαλία και Φιλανδία. 27 εμπειρογνώμονες τοποθετήθηκαν και ήρθαμε σε επαφή με πολλούς άλλους ακόμα. Αυτές οι συνεντεύξεις συμπληρώθηκαν από εξέταση των διαφόρων εκθέσεων, διαφόρων εγγράφων. Θέλαμε όλα τα συμφέροντα να συμμετάσχουν. Να λεφθούν υπόψη διάφορες απόψεις και ενδιαφερόμενοι από τη βιομηχανία, οικειό, κυβερνητικούς φορείς και πανεπιστημιακούς κύκλους. Δοθέντος του καθήκοντος αυτού και του χρόνου ε, δεν είναι αντιπροσωπευτικό το έγγραφο πλευρά στατιστική. Ζητήσαμε λοιπόν στην υπηρεσία κοινοβουλευτική έρευνα του εμπειρογνώμε μα πούν σε ποιο βαθμό οι στόχοι τη οδηγία έχουν εκπληρωθεί. Κυρίω όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα και εμπόδια που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τη οδηγία, Πώ η οδηγία επηρεάζει άλλε πολιτικέ και νομοθεσία. Πώ η οδηγία συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και πού μπορεί ε, να επιδέχεται βελτιώσεων. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι τη οδηγία. Τι λέει η οδηγία. Θέλει να πετύχει υψηλό επίπεδο προστασία του περιβάλλοντο. Θέλει να μειώσει τον αντίκτυπο των περιβάλλων των διαφόρων προϊόντων που μπορει να επιδεχεται βελτιωσεων ποιοι ειναι οι βασικοι στοχοι τη οδηγια τι λεει η οδηγια θελει να πετυχει υψηλο επιπεδο προστασιας του περιβαλλοντος θελει να μειωσει τον αντικτυπο του περιβαλλον των διαφορων προιοντων που σχετιζονται με την ενέργεια. Στην ίδια παράγραφο. Λέει ότι η βελτίωση αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας συμβάλλει στον ασφαλή εφοδιασμό ενέργεια και στη μείωση της ζήτησης ε, για φυσικούς πόρους. Τα διάφορα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια, ποια είναι αυτά. Αυτά που χρησιμοποιούν ενέργεια ή προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια, αλλά έχουν αντίκτυπο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργεια. Παραδείγματο χάρη, προϊόντα μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση σε κτίρια. Εν γέννη, όλοι εξέφρασαν την άποψη ότι η οδηγία ήταν επιτυχέστατη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Όμω συμφωνούν ότι δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα η αποτελεσματική των πόρων εντός των κανονισμών περί προϊόντων πέραν της συνολική αποδόσεως. Άρα η αποδοτικότητα των υλικών. Αυτό σχετίζεται με το τέταρτο θέμα που αφορά την κυκλική οικονομία. Συζητώντας το θέμα αυτό της χρήσης των υλικών και των υλικών που χρησιμοποιούνται υπήρχαν αποκλίνουσες απόψεις. Δύο επιχειρήματα προευλήθησαν. Πρέπει οι απαιτήσει για τελικά να τονιστούν μετά είπαν άλλοι ότι υπάρχουν προβλήματα, φραγμοί για τη χρήση των υλικών. Λοιπόν, μας είπαν οι εμπλεκόμενοι φορείς και ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχουν όρια όσον αφορά τις απαιτήσει για ενεργειακή απόδοση ε, λόγω περίπλοκου χαρακτήρα των μέτρων. Η πλειοψηφία πιστεύει επίσης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι απαιτήσει για την ε, ενεργειακή απόδοση των υλικών και απαιτήσει όμως που μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι μέτρησιμες από τις αρμόδιες αρχές. Τρίτη θέση, πιο φιλόδοξη. Λίγοι το έσπρωξαν αυτό. Είπαν ότι τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια μπορεί να επεκταθούν και να μπουν και άλλα προϊόντα που δεν είναι βαθμολογημένα ενεργειακά όπως είναι τα έπιπλα, βασικά εμπόδια. Όλοι είπαν ότι είναι μακρά η ρυθμιστική ε, διαδικασία και ο τη αγορά. Χρονοβόρες οι διαδικασίες για να ο κανονισμό. Κυρίω για προϊόντα που είναι πολύ προθυμένα τεχνολογικά. Και έτσι χάνουμε οικονομίες ενέργειας και δεν πετυχαίνουμε επαρκείς στόχους. Υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει και έλλειψη στελέχωσης, ε, έλλειψη προσωπικού, διότι διερκώς διευρύνει το τομέας. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι η εποπτεία της αγοράς δεν πηγαίνει καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως είναι σημαντικός παράγον για να πετύχει οδηγία. 10 με 25% των προϊόντων στην αγορά που ρυθμίζονται από την οδηγία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσει για οικολογικό σχεδιασμό. Γιατί? Υπάρχουν πολύ λίγοι πόροι στα κρατη Κάθε χώρα κάνει δικέ τη δοκιμέ για τα προϊόντα. Κάτι δαπανηρό. Απαιτεί τεχνογνωσία και εγκαταστάσει δοκιμών. Άλλο. Έλλειψη σαφών προδιαγραφών και προτύπων. Έλλειψη προσανατολισμών για μεθόδους ελέγχου και βαθμολόγησης για να δούμε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση ε, με τον κανονισμό όσον αφορά τις επαιτήσεις περί χρησιμοποιημένων ε, υλικών. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Οι συστάσεις που βλέπετε. Να συνεχίσουμε να συμπεριλαμβάνουν περισσότερα προϊόντα που σχετίζουν ενέργεια να αξιολογηθεί η δυνατότητα να ρυθμίζουμε προϊόντα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια, να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι εφικτό να ρυθμίζουμε προϊόντα όσον αφορά τι απαιτήσει για αποδοτικότητα των υλικών, χρονοδιαγράμματα για συμφωνία του κανονισμού και να τηρείται το χρονοδιάγραμμα, καλείται το συντονισμό μεταξύ εθνικών αρχών υποπτία τη αγορά και χρειάζονται συμπεφωνημένοι προσανατολισμοί για τον έλεγχο και τι δοκιμέ των προϊόντων και τι, πρέπει, τι μήτρα πρέπει να χρησιμοποιούν οι διάφορε αρμόδιε αρχέ που ελέγχουν την αγορά για να κρίνουν τα διάφορα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χαβιέ Μπουράνη από την ε, Βαρκελόνη, την Καταλωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εφαρμογή του οδηγία μέσω του σχετικού κανονισμού έχει ε, επίπτωση στην, στον κύκλο ζωής. related products become more efficient, becomes more relevant. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο τα θέματα όσον αφορά τον κύκλο ζωής που θα πρέπει ε, να ε, δώσει, να οδηγήσει σε βελτίωση και των, προ, των πρώτων και της παραγωγής αλλά και της διαχείρισης του κύκλου ε, ζωής. Όσο πιο πράσινες είναι οι ενέργειες, τόσο καλύτερος θα είναι ο κύκλος ζωής. Ο ενεργειακός κανονισμός θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να συμπεριλάβει και την ιδέα της, ε, της ε, περιβαλλοντικής προληπτικής αρχής που θα ακολουθήσει το προϊόν από τη δημιουργία μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής και με τον τρόπο αυτό να προχωρήσει και η κυκλική οικονομία. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως το στοιχείο αυτό ε, να ληφθεί υπόψη στα πρώτα στάδια σχεδιασμού του προϊόντος ε, και πρέπει οπωσδήποτε να ε, είναι σωστός ο σχεδιασμός έτσι ώστε να μπορέσει να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Εδώ σας βλέπω διάφορους λαμπτήρες όπως βλέπετε. Design variability. OLEDs ε, εδώ όμως ε, δεν είναι πράγματα για πέταμα γιατί περιλαμβάνουν ε, πολλά, πολλές σημαντικές πρώτες ύλες. Το ξέρουν αυτό οι επιχειρήσεις, αλλά ο σχεδιασμός είναι τέτοιος που η ανάκτηση των σπανίων υλικών οικονομικά δεν γίνεται και πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως τα προϊόντα αυτά, όπως αυτοί οι λαμπτήρες, δεν είναι πάρα πολύ εύκολοι στην ανακύκλωσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οπωσδήποτε πιο αποτελεσματικοί οι λαμπτήρες, αλλά οπωσδήποτε να, από την ε, στιγμή της σύλληψής τους και του σχεδιασμού τους ε, να ε, σχεδιαστούν με τρόπο ώστε στο τέλος της ζωής τους να μπορούν γρήγορα και εύκολα να ανακτηθούν τα σημαντικά υλικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ε, ουσιαστική κυκλική οικονομία. Εμείς αναλύσαμε έξι ειδών προϊόντα. Ε, αυτά τα προϊόντα έχουν τελείως διαφορετικό καθεστώς, βλέπετε με διαφορετικά ε, χρώματα, είτε ανήκουν σε διαφορετικούς ε, κανονισμούς. έχουμε ας πούμε τηλεοράσεις, έχουμε σκούπες ηλεκτρικές, έχουμε ψυγεία, έχουμε θερμοσύφωνα, θερμαντήρες νερού κτλ. Το κεντρικό μας μήνυμα είναι ότι βρισκόμαστε ήδη στον καλό, στο σωστό δρόμο, γιατί δύο από, τα έξι, δύο από τις έξι ομάδες προϊόντων περιλαμβάνουν ε, κάποιον ε, ε, ενεργειακό, κάποια ενεργειακή επισήμανση ας πούμε και ταξινόμηση. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε ανάλυση της χρήσης, τη φάση της χρήσης. Αλλά μονάχα οι λαμπύρες ε, και οι, ε, και οι σκούπες ηλεκτρικές που βλέπετε αριστερά στην εικόνα ε, έχουν κάποια αναφορά στον κύκλο ζωής και για τον τρόπο με τον οποίο θα ανακυκλωθούν στο τέλος της ζωής του. Το δεύτερο μήνυμά μας είναι ότι για όλα ε, τα προϊόντα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ανάλυση όσον αφορά θέματα ε, που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, δηλαδή ε, δυνατότητα ανακύκλωσης, επανάχρησης, επανάχρησης ορισμένων στοιχείων, επιδιόρθωσης κλπ. Θα πρέπει επομένως οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τεχνικές προδιαγραφές ε, ήδη από τα πρώτα στάδια σύλληψης και σχεδιασμού του προϊόντος. Τρίτο μας μήνυμα είναι ότι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να, ευθυγραμμίζεται με άλλους στόχους και άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία. Έχουμε ας πούμε την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, έχουμε την οδηγία για την ε, ανακύκλωση των αποβλήτων κλπ μέσα από μία συνδυασμένη αντιμετώπιση θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην κυκλική οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω αναφερόμενα στην έκθεσή μου ή θα έχουμε ρωταπαντήσεις με τους δύο εμπειρογνώμονες. Ίσως καλύτερα να ξεκινήσω άμεσα. Πιο εύκολο θα είναι. Σκεφτόμουν να μας πείτε αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά την παρουσίαση που έγινε. Την έκθεση θέλετε να αναφέρετε. Είναι κοινή συζήτηση μαζί με την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράμπη και τον κύριο Καμπαρέλ για αυτή την παρουσίαση που ήταν πληρέστατη και που σίγουρα είναι πολύ καθησυχαστή και στον αφορά τη δική μου έκθεση. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η μελέτη αποτελούσε τη βάση επί της οποίας ε, στήριξα την έκθεσή μου εν μέρη, τις διαπιστώσεις μου και τις προτάσεις μου. Και συμφωνούμε όσον αφορά τα βασικά στοιχεία. Τίθεται το θέμα της οδηγίας ε, περί της οικολογικής αυτής ε, σύλληψης ιδιασμού ε, μας παρουσιάστηκαν διάφορες φωτογραφίες παρουσιάζοντα το θέμα που καλύπτουν διάφορα προϊόντα τα οποία συνδέονται με την ενέργεια, οικιακέ συσκευές, τηλεοράσει, οθόνε θερμαστρές κλπ. Ε, Βραστήρε, ε, ηλιακοί συσσωρευτές κλπ. Η οδηγία για, την, για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι κάτι παραπάνω από ένα εξαιρετικό εργαλείο. Δεν είπαμε αρκετά για αυτήν. Νομίζω ότι έχουμε επίγνωση αυτού όταν μιλάμε για ευαισθητοποίηση των πολιτών, πόρο απέχουμε από το στόχο. Είναι σημαντικό αυτό. Επανέρχομαι λοιπόν στο εργαλείο που αποτελεί αυτή η οδηγία, ένα πραγματικό πυλώνα προς την ενεργειακή αποδοτικότητα της κυκλικής οικονομίας. Θα ήθελα να παραθέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διευκρινίζει ότι αυτή η οδηγία για, την, για τον οικολογικό σχεδιασμό και ο κανονισμός για την ιδιοθεσία για, το, για την οικολογική σήμανση ε, μας οδηγούν σε, στους μισούς στόχους που έχουμε θέσει για το 2020 για την εξοικονόμηση ενεργείας. Τεράστιο αυτό. Αυτό δείχνει τι δουλειά κάνουμε. Αυτή η διαπίστωση επανειλημμένα αναφέρθηκε από όλου του παρεμβαίνοντε στον κοιλό τραπέζι που διοργάνωσα με, με τη Μισελ Ριβαζή, εισηγήτρια για γνωμοδότη τη Επιτροπή ΣΥΤΡΕ, στι 23 Ιανουαρίου εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, έγινε αυτή η συζήτηση. Ε, Λοιπόν, πάντα με τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ετικετοθεσία και όλη η πολιτική σχεδιασμού 177 εκατομμύρια ισοδύναμων τόνους πετρελαίου ε, το χρόνο ήταν η οικονομία σε ενέργεια και η κατανάλωση της ενέργειας αντιστοιχεί στη σημερινή ε, κατανάλωση της Ιταλίας σε ένα χρόνο. Ε, λοιπόν, στα πιο καθημερινά για τους καταναλωτές μας περίπου αυτό τη στοιχή, 490 ευρώ ανανοικοκυριό το χρόνο όσον αφορά τους λογαριασμούς ενέργειας. Ε, δεν αμελείται αυτό. Είναι μια επιτυχία που επιβεβαιώνει θα έλεγα επιβεβαιώνεται από τις Βρετανικές Αρχές. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2015 που συνεπεράνε ότι κάθε λίρα που επενδύεται στο οικολογικό σχεδιασμό έδινε, έδινε 3,8 λίρε στη Βρετανική οικονομία. Άρα είναι αποδοτικέ αυτέ οι προσεγγίσεις. Είναι όταν ξέρουμε σε ποιο βαθμό από αυτά διαβάσαμε και στην ε, προεκλογική εκστρατεία την προηγούμενη στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την οδηγία τη συγκεκριμένη. Είναι ηρωνικό αυτό. Υπάρχουν αλήθειες που είναι καλό να υπενθυμίζονται εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το τοπίο υπάρχουν και κάποια προβλήματα βέβαια διότι ε, διάφορες επικρίσεις ακούστηκαν. Τις ακούσαμε και εδώ. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις, τους αργούς ρυθμούς λήψεως αποφάσεων. Το 2004 στην επεξεργασία της πρώτης οδηγίας πλαίσιο, ήμουν τότε εισηγήτρια, καταφέραμε με μια με τις ομάδες της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ηγητές στο Κοινοβούλιο, Πίτερ Λίζερ και τον Κλό Τούρμες, καταφέραμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα φανταστικό εργαλείο, το Φόρουμ Διαβούλευσης. Εκεί συμμετέχουν οι ΜΚΟ, εκπρόσωποι βιομηχανία και εθνικοί εμπειρογνώμονες, οι stakeholders Θέλαμε να δούμε κατά πόσο ένα συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να υποβάλλεται σε ένα μέτρο οικολογικού σχεδιασμού, ετικετοθεσία ενεργειακή ή όχι ε, σε μια ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους, βάσει αυτής της αναλύσεως κόστους-οφέλους. Αυτή η διαδικασία είναι μακροσκελέστατη, πάρα πολύ αργή, δεν δίνει τα απαραίτητα χέγγια στους παραγωγούς και γι' αυτό επιμένω στην παράγραφο 4 συν 5 και 6 τη εκθέσεω συγγνώμη, όσον αφορά την υποχρέωση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει την κατάσταση, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστέ θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται και να τηρούν τι προκαθορισμένε συγκεκριμένε προθεσμίε. Είναι πολύ βασικό η στρατηγική για να έχουμε και θεμητό ανταγωνισμό σε σχέση με αυτά που έρχονται απ' έξω, από μη Ευρωπαίου παραγωγού. Λοιπόν, ε, αλλάζει και ο προσανατολισμό όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Κατάιν έδωσε κάποιες απαντήσεις σε πολλοί ερωτήσεις που ετέθησαν και θεωρώ ότι αυτά που ακούσαμε ήταν ενθαρρυντικά, κυρίως όσον αφορά ότι δεν πρέπει να εστιαζόμαστε αποκλειστικά επί της ενεργειακής απόδοσης. Ο Επίτροπος ε, είπε και παραθέτω η χρήση των πόρων και η ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων. Και εγώ συμφωνώ προφανώς, είναι σημαντικά σημεία, κρίσιμα θα έλεγα, που αναφέρονται στην έκθεσή μου και αφορούν το συσχετισμό με τρίτο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που αναφέρθηκε του εμπειρογνώμονε. Δηλαδή, ποιο είναι ο στόχο μα, να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την εποπτεία των αγορών. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να περάσουμε από μια οικονομία και μια λογική τη εξοικονόμηση ενέργεια, να πάμε σε εξοικονόμηση των πόρων. Αποτελεσματικότητα των πόρων αυτή εν μέρει έχει ενταχθεί στο σχέδιο εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φτάνει μέχρι το 2019 και αυτό για μια σειρά προϊόντων, ε, τηλεοράσεις, ε, σκούπες κλπ. Ε, δεν βασιζόμαστε πάντα στα ίδια κριτήρια. Καμιά φορά έχουμε τη βελτίωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος, είναι κάτι που μελετάτε. Άλλες φορές τονίζεται το τέλος ζωής, η πτυχή της ανακύκλωσης του προϊόντος που μελετάτε, η δυνατότητα να γίνει αποσύνθεση του αγαθού στα διάφορα συστατικά του. Όπω είναι τα κινητά τηλέφωνα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια κατά περίπτωση προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείτε, είναι καλή. Μετά και κάτι άλλο, το οποίο ομόφωνα στηρίχτηκε και απαιτήθηκε από του ενδιαφερόμενου φορεί τη συζητήση των κ. Τραπέζη του περασμένου μηνό, Το θέμα τη εποπτεία των αγορών και των διαφορών που υπάρχουν, αποκλήσεων που υπάρχουν, περιπτώσει, μη εποπτεία και τα αριθμητικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. 10 με 25% των προϊόντων που ρυθμίζονται από την υγεία δεν ε, συμμορφούνται. Ένα προϊόν στα τέσσερα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, έχω προτάσεις και συστάσεις στην έκθεσή μου που αφιερώνονται σε αυτή την πτυχή στις παραγράφους 11 μέχρι 13. Θα βελτιωθούν και προτάσεις των συναδέλφων. Θα επεκταθεί η βάση δεδομένων της Ευρώπης όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς ή σε SMS που αποκαλείται και όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων ε, θα μπορούσε να επεκταθεί επίσης και στις επιδόσεις της περιβαλλοντικές των προϊόντων. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνω. Ε, και άλλα δύο επικέρα θέματα. Ε, λοιπόν, τα κινητά τηλέφωνα θα μπουν στο σχέδιο εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο, η πρώιμη γύρανση, αν θέλετε, και που απαρχαιώνονται τα προϊόντα πολύ γρήγορα. Ε, για την ώρα δεν υπάρχουν σχετικά ευρωπαϊκά μέτρα. Είναι εύκολο βλέποντα ότι είναι ταχύτατη η εξέλιξη, στιγμία η εξέλιξη θα λέγα της τεχνολογίας. Ε, δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε τον οικολογικό σχεδιασμό λόγω των ταχυτάτων τεχνολογικών εξελίξεων ε, ας πούμε έχουμε τις ολοκληρωμένες, έχουμε τις μπαταρίες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν και πετάμε τις συσκευές και τα τηλέφωνα παραδείγματος χάρη. Λοιπόν στην παράγραφο 10 ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει τα κινητά τηλέφωνα αυτά στο σχέδιο εργασιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και είναι μια από τις ερωτήσεις μου προς ε, υπευθύνους, τους εμπειρογνώμονες. Τι σκέφτονται γι' αυτό. Ε, πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα όσον αφορά ε, τον πρώιμη λήξη κύκλου ζωής. Λοιπόν, στην έκθεση του Ιράν αναφερόμαστε σε κάτι άλλο. Υιοθετήσαμε πέρσι τον Ιούλιο, στην παράγραφο 8, τα συστήματα ετικετοθεσίας επίσης ε, δηλαδή διάρκεια ζωής πώς θα αναφέρεται στην ετικέτα στον καταναλωτή ε, η διάρκεια ζωής του προϊόντος που αγοράζει είναι μια έξοχη ιδέα η οποία θα πρέπει να εμφανίζεται ε, στην τελική μας έκθεση. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you very much. Now I Ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τους κοιόδους τώρα. Άμα θέλετε μπορείτε να σχολιάσετε και την έκθεση και το σχέδιο έκθεσης της ε, κυρίας Δρύς, ο κύριος Κάμπους. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το IPRS για την ε, εργασία που έκανε γιατί πραγματικά μα έδωσε πολύτιμα στοιχεία για, την κοινοβουλευτική μας, ε, για το κοινοβουλευτικό μα έργο. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το έργο τη ε, και για τι προσπάθειε που έχει καταβάλει έτσι ώστε το κείμενο να είναι όσο γίνεται πιο συνενετικό και μάλιστα εξ αρχής. Συμφωνούμε, συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία τη κυρία Ρίσα κυρίω εκεί που αναφέρει την ανάγκη να αλλάξουμε την αντίληψη του οικολογικού σχεδιασμού. Ε, θα πρέπει η ευρωπαϊκή οικονομία να προχωρήσει και να γίνει κυκλική οικονομία και λέμε ότι πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν λειτουργούν αυτές οι λύσεις που είχαμε μέχρι τώρα και πρέπει να βρούμε καινούριε. Θα πρέπει να δουλέψουμε και με τους χρήστες αλλά οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να εργαστούμε χέρι με χέρι και με την βιομηχανία που αυτή θα πρέπει να πραγματοποιήσει υλοποιήσει τούτη την αλλαγή συζητούμε, ε, ασχολούμαστε με θέματα τα οποία αφορούν τους χρήστες, εμάς που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα ε, αυτά τα ε, προϊόντα και επομένως η, σωστή χρήση της, του οικονομικού σχεδιασμού μπορεί να μας εξοικονομήσει πολλά χρήματα κάθε χρόνο. Θα πρέπει επομένως να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα βήματα τα οποία αναλαμβάνουμε καθώς επίσης και για το όφελος που μπορούμε να έχουμε. Ένα άλλο σημείο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να υποραμιστεί είναι ότι η κυκλική οικονομία είναι εγκάρσια διαδικασία. Ε, η συγγήτρια αναφέρθηκε στην παρουσία του Αντιπροέδρου Κατάινεν την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμα και το γεγονό το ίδιο ότι ήρθε ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα μιλήσει για τα θέματα αυτά ε, δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά και ότι πραγματικά δεν μπορούμε, ε, δεν μπορούμε να δούμε την ε, κυκλική οικονομία και το τον ε, οικολογικό σχεδιασμό σαν ένα ενιαίο στοιχείο. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, θα πρέπει και το οικολογικό σχεδιασμό και την κυκλική οικονομία να τις δούμε με φιλοδοξία, μέσα σε φιλόδοξα σχέδια οπωσδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να περιορίσουμε τον οικολογικό σχεδιασμό στην εξοικονομία εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πρέπει να ξαναδούμε την δυνατότητα ε, χρήσης, επανάχρησης στοιχείων, ανάκτησης και επανάκτησης ε, πρώτων υλών, διαεύρυνση και επιμήκυνση του κύκλου ζωής κλπ. Και οπωσδήποτε δεν πρέπει ούτε μισό βήμα να κάνουμε προς τα πίσω. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε ακόμα. Δεν είναι δυνατόν ε, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσουν πρόσκομα στην πρόθεση της, ε, του οικολογικού σχεδιασμού και εδώ κατά την έννοια αυτή ε, θα ρωτήσω και εγώ όπως και η συγγήτρια ποια ε, ιδέα έχετε, πώ πώς αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία αυτή τα κινητά τηλέφωνα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Τελειώνοντας να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την εισηγήτρια για την έκθεση που παρουσίασε ε, και συμφωνούμε με τα περισσότερα από όσα αναφέρει το κείμενό της. Θα θελήσουμε βεβαίως να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο μέσα από τροπολογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταλή, εξ ονόματος κυρίου Παολούτσι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω την κυρία Ρίσε για το προσχέδιο έκθεσης το οποίο μας έχει υποβάλει. Να ευχαριστήσω και το EPRS για την μελέτη που έκανε και ευχαριστούμε και την autonoma της barcelona που μας έκανε την παρουσίαση σήμερα. Ο Μάσιμο Παολούτσι, ο σκιώδης ε, θεωρεί ότι η έκθεση αποτελεί καλή βάση για συζήτηση γιατί ήδη περιλαμβάνει πολλέ πολλές θετικές ε, προτάσεις όσον αφορά ε, την εφαρμογή του, κανο, του τη, της οδηγίας ε, για τον οικολογικό σχεδιασμό. Προτίθεται να υποβάλει κάποιες τροπολογίες έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η έκθεση αυτή. Ε, θα αφορούν δε την εποπτεία της αγοράς γιατί πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και επίσης ε, θα πρέπει να κοινοποιούνται όλες ε, οι, όλοι οι έλεγχοι συμμόρφωσης ε, που γίνονται σε μια χώρα μέλος και να δημιουργηθεί ενδεχομένως ε, μια νέα ε, υπηρεσία επιτήρησης αγοράς. Ε, δεύτερο σημείο, ισχυρότερη επιτήρηση η οποία θα πρέπει να βασίζεται και σε εθελούσιες εθελοντικές συμφωνίες για εισαγόμενα προϊόντα. Τρίτο σημείο, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα αφενός στον οικολογικό σχεδιασμό και αφετέρου την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν επιθεωρήσεις όσον αφορά ε, την ενεργειακή απόδοση, όσον αφορά την ε, εφαρμογή του κανονισμού για, την, ε, για τα δομικά υλικά και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί ο, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αρχή των ελάχιστων ε, ανακτήσιμων πρώτων υλών καθώς επίσης και για τη δυνατότητα ανάκτησης σπανίων μετάλλων. Επίσης ε, το σημείο που αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει σε μια πραγματική ενιαία αγορά. Τέταρτο, ε, πέμπτο, συγγνώμη, πλήρη συνεργασία με την κυρία Ρίσε καθώς επίσης και με τους άλλους σκιώδεις σύγητες έτσι ώστε να δούμε το θέμα από όλες τις πλευρές του. Ο κύριος Πιακα, εξ ονόματος της κυρίας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτριά μας για την παρουσίαση που έκανε, το σχέδιο εκθέσεως και εν ονόματι της κυρίας Βυσσινιέσκα. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα σχόλια που έχει όσον αφορά αυτό το σχέδιο εκθέσεως. Εδώ αναφερόμαστε στην εφαρμογή της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασμού και αυτό το κείμενο το κρίνουμε ε, θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει τους στόχους της όσον αφορά το κλίμα και μπορεί να επιτρέψει και σημαντικές ε, μειώσεις ε, κατανάλωσης ενέργειας στους Ευρωπαίους πολίτες. Το κείμενο που προτείνεται είναι καλό κείμενο, το ψήφισμα, όσον αφορά την κυκλική οικονομία. Τα προϊόντα που σχεδιάζονται σήμερα θα πρέπει να είναι βιώσιμα και δεν θα πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια με την πρώτη βλάβη τους. Θα πρέπει οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν ότι μπορούν να επιδιορθώνονται αυτές οι συσκευές και έτσι η διάρκεια χρήσεως αυτών να είναι η πλέον μακροχρόνια όσο πιο μακροχρόνια μπορεί να είναι. Είναι σημαντικό να εξετάζεται και ενεργειακή απόδοση αυτό είναι σημαντικότατο στοιχείο. Είναι η πιο σημαντική απέτηση όσον αφορά τα νέα προϊόντα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αν έχουμε νέες απαιτήσει, αυτές θα πρέπει να δικαιολογούνται τεχνολογικώς και θα πρέπει τα μέτρα αυτά να είναι εφαρμόσιμα. Θα πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην αυξάνεται πολύ το κόστος παραγωγής, να μπορεί να είναι ανταγωνιστικέ οι εταιρείε. Η οδηγία αυτή για τον οικολογικό σχεδιασμό θα πρέπει να βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε και όλες τις προτινόμενες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση, λέει η κυρία Όκεν. Είναι πολύ καλό να συζητούμε με αυτόν τον τρόπο τα ζητήματα. Πάμε πίσω στην προεκλογική εκστρατεία. Είχαμε προβλήματα στις χώρες μας, διότι ο κόσμος τότε δεν καταλάβαινε περί τίνος επρόκειτο όσον αφορά την οδηγία έλεγαν ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις καφετιέρες μας και με τις συλλεκτικές μας κούπες. Τι θέλει. Ε, Ήταν σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της οδηγίας και πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Το πιο σημαντικό της εκθέσεως είναι ότι μπορούμε να υπογραμμίσουμε την επιτυχία της οδηγίας και ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ε, χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου, χρειαζόμαστε καλύτερες φάσεις εφαρμογής των μέτρων και όπως υπόθηκε και από την κυρία Ρης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι στόχοι θα καλύπτουν και την αποδοτική χρήση των πόρων. Και θυμάμαι, όταν ήμουν κάπως νεότερη πολιτικός στο Κοινοβούλιο της Δανίας, τότε λοιπόν συζητούσαμε τη νέα τεχνολογία της πληροφορικής και τότε μας έλεγαν ότι σε λίγο θα έχετε τα μηχανήματα ε, θα μένουν τα μηχανήματα και το μόνο που θα αλλάζει κανείς θα είναι το λογισμικό. Θα ήταν υπέροχο αν αυτό ίσχυε. Δηλαδή να αγόραζε κανείς το μηχάνημα και μετά να βελτιώνει μόνο το λογισμικό. Αλλά τελικά αυτό που ξεπερνιέται πιο γρήγορα είναι το, το μηχάνημα και το λογισμικό, όπως βλέπουμε τα κινητά, ε, που έχουν ε, ένα, μια, ένα, ε, μια λήξη κύκλου ζωής. Όταν κάνεις αναβάθμιση του λογισμικού βελτιώνεται η αποδοτικότητα, αλλά αμέσως μετά πρέπει να αλλάξει τη συσκευή. Παλιά θεωρούσαμε ότι θα μπορούμε να ανακυκλώνουμε περισσότερο. Εκεί δεν έχει δοθεί δεύτερη προσοχή, πολύ λίγη προσοχή δόθηκε στην ανακύκλωση. Δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ. Αυτό είναι εκπληκτικό βλέποντας το πώς κάνουμε διαλογή των αποβλήτων και πόσο λίγη ανακύκλωση γίνεται παρά τη διαλογή και πόσο λίγη ζήτηση υπάρχει. Χαίρομαι που εδώ δίνουμε την κατάλληλη προσοχή στο θέμα της ανακύκλωσης. θα πρέπει να αποφύγουμε να μην διευρύνουμε υπερβολικά το πεδίο. Διότι ίσως τελικά το παρακάνουμε και ίσως να μην λειτουργεί στο σύστημα. Θα μας λένε μετά ότι επιβάλλουμε απαιτήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κανείς ο απλός άνθρωπος δεν μπορεί να εφαρμόσει τις απαιτήσει και ότι στριμώχνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που λένε κάθε φορά οι άνθρωποι όποτε συζητείται αυτό το θέμα. Λοιπόν αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Μην επεκταθούμε υπερβολικά. Οι περισσότεροι όμω συμφωνούν με τις γενικές γραμμές. Ευχαριστώ. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση που έγινε της μελέτης και ευχαριστώ και την εισηγήτρια έξοχη γνωμοδότηση την οποία παρουσίασε ε, και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι τα ωφέλη αυτής της οδηγίας είναι προφανή τα θετικά της στοιχεία αναμφισβήτητα πετύχαμε οικονομίες όσον αφορά τη χρήση της πρωτογενούς ενέργειας αλλά αποφύγαμε να εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακο στο περιβάλλον, ε, κάναμε και οικονομίες για τους καταναλωτές. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε, να βελτιώσουμε πάρα πολύ και να αυξήσουμε τις, ε, τη φιλοδοξία του νομοθετικού κειμένου. Και το λέω επίσης επειδή συμφωνώ με αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι, ότι δεν θα πρέπει μόνο να μιλάμε για ενεργειακή απόδοση των προϊόντων, αλλά θα πρέπει και είναι επιτακτική ανάγκη να μιλήσουμε και για την αποδότητα των υλικών, για του ε, πόρου, για τι πηγέ, για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα. Ξέρουμε πολύ καλά πως από την αρχική φάση του σχεδιασμού μπορεί κανείς να καθορίσει ε, πόσο θα επηρεάσει το περιβάλλον ένα προϊόν συνεπώς τι γίνεται με τη ρήπανση κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής ε, του ίδιου του προϊόντος. Είναι θεμελιώδες να γίνεται σωστός σχεδιασμός. Για να γίνει αυτό, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε από άλλου συναδέλφου. Είναι απαραίτητο και εδώ επιτακτική ανάγκη, θα έλεγα, να μιλάμε για τη διάρκεια των προϊόντων, να μιλάμε για ανάκτηση, επανήχρηση, χρήση των διαφόρων ανταλλακτικών και των διαφόρων κομματιών του μηχανήματος ε, θα έχει υποχρεωτικές απαιτήσεις το επιβάλλει όσον αφορά τη δυνατότητα να έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής τα προϊόντα και να χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Έγινε μια μελέτη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα της ΕΠΑ, της ε, υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΕΠΑ, που λέει ότι για 10.000 τόνους αποβλήτων δημιουργείται με θέσει εργασία για την κάψη έξι θέσει εργασία ε, στη χώρα αποβλήτων ε, και στην ανακύκλωση έξι θέσει και 294 θέσει εργασία στην όλη ε, γραμμή ανάκτησης, ανακύκλωσης και επιδιόρθωσης των προϊόντων. Είναι μια δυνατότητα να το δεχτούμε αυτό και για την αντίκτυπο που έχει για θέσεις απασχόλησης. Δημιουργεί και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Πότε μπορούμε να δούμε κάποιο δείκτη όπως ε, του άνθρακα, ένα ίχνος ε, για τα προϊόντα όπως είναι και το ίχνος άνθρακα. Είναι σημαντικό αυτό για να ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτές και πότε θα μπορέσουμε να δούμε και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποιο κίνητρο κάποια υποστήριξη για να περάσουμε από οικονομία που εδράζεται επί κατοχής του προϊόντος, επί μέση οικονομίας που βασίζεται επί των υπηρεσιών. Λοιπόν, οπότε είναι κερδοφόρα για όλους. Κερδίζουν εκεί καταναλωτές που έχουν προϊόντα που λειτουργούν όλο και πιο περισσότερο χρονικό διάστημα και για εκείνους που παρέχουν τι υπηρεσίε που έχουν συμφέρον να λειτουργούν καλά με την πάροδο του χρόνου τα προϊόντα και να διατηρούν αναλύωτα τα χαρακτηριστικά τους. Ε, ευχαριστώ την συγκέντρια για τη δουλειά που έκανε και μόλι ελπίζουμε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τη Φρεντερή Τα σχόλια της, τα επιχειρήματά της ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, όμως αυτή η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό επικεντρώνεται στην ε, μείωση κατανάλωση ενέργειας κατά τη ε, διάρκεια χρήσης των προϊόντων και δεν επικεντρώνεται αρκετά κατά τη γνώμη μου στο δυναμικό εξοικονόμησης μέσα στην κυκλική οικονομία διότι ε, η έννοια του κύκλου ζωής ε, έχει κύρια σημασία για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για να αυξήσουμε την δυνατότητα επαναχρησιμοποίηση. Οπότε χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση να παρατείνουμε ε, τον ε, κύκλο ζωής ε, των μηχανών και των υλικών που χρησιμοποιούμε. Αυτό για την ανακύκλωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από αυτό πρέπει να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γι' αυτό χρειάζεται μια κατά περίπτωση δεόντως περιστατωμένη προσέγγιση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και στις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστούμε. Ριβαζή. Ήμουνα εισηγήτρια ε, για, στην Ήτρε για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ τη Φρεντερή Κρίς ε, για τη δουλειά που έκανε και για τη συνεργασία των σκιωδών. Ε, λοιπόν, στην Ήτρε, και πανέρχομαι τώρα σε αυτά που μόλις μας είπε η κυρία Γκροστέτ, ε, μιλήσαμε για την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής κατανάλωσης. Ναι, αυτό είναι θετικό γιατί ασχοληθήκαμε με το θέμα της ετικετοθεσίας. Αλλά πέρα από αυτό χρειαζόμαστε αποτελεσματικά ε, υλικά για να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε και κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού για να εξοικονομήσουμε πόρους για την κυκλική οικονομία και για την υγεία. Ε, και είναι περίεργο που δεν μιλάμε ε, για το θέμα της υγείας ε, όταν πραγματευόμαστε τον οικολογικό σχεδιασμό σε αυτή την Επιτροπή. Λοιπόν, η βιωσιμότητα των υλικών πρέπει να είναι βιώσιμη τελικά. Δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τελικά μία χρήση, να παρατείνουμε τον κύκλο χρήση. Γιατί αυτό είναι πολύ πιο εύκολο σε σχέση με την προγραμματισμένη το προγραμματισμένο τέλος ε, ζωής ενός προϊόντος. Ε, δηλαδή, αν πρέπει, καταλαβαίνετε, να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας αδύναμος λίγο στην ε, παρασκε... κατά την κατασκευή ενός προϊόντος, ε, καταλαβαίνετε τι δυσκολίε συνεπάγεται αυτό, όπως έγινε με τα αυτοκίνητα και τις εκπομπές που τελικά καταλήξαν στο ότι έφυγε ένα ε, λογισμικό. Ε, πέρα από αυτό, ε, η έννοια του ανακυκλώσιμου, για κοιτάξτε γύρω σας, ε, δεν είναι αδιανόητο που συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε προϊόντα που δεν είναι 100% ανακυκλώσιμα, πλαστικά. Πλαστικά συνεχίζουν να παράγουν πλαστικά που δεν είναι 100% ανακυκλώσιμα και συσσωρεύονται τα απόβλητα. Και εφόσον έχουμε εδώ πέρα και εξωτερικούς συμβούλους και επαϊόντες, θα ήθελα την άποψή σας, τι να κάνουμε για να πιέσουμε πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα τα προϊόντα γιατί θα ε, ε, ε, μας κατακλείσουν τόνοι βουνά απορριμμάτων αποβλήτων. Ε, τώρα, όταν βλέπω το 96% της, παρασκευ... της κατασκευής γίνεται στην Κίνα, τι κάνει η Ευρώπη. Εγώ είμαι οικολόγος. Είτε μιλάμε για την ελληνική ενέργεια, φωτοβολταϊκή ενέργεια κινητά, όλα ε, είναι ε, σπάνιες γιές. Και λοιπόν τι κάνει η Ευρώπη. Γιατί έχει αυτό το μερίδιο λέοντος η Κίνα. Ε, έχουμε πει στους ενδοκρινικούς διαταράκτες και και τα πολυοργανικά θεκτικά υλικά ε, Όντω θα πρέπει να εντείνουμε την ε, εποπτεία της αγοράς και θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να υπάρχουν και τα μέσα ελέγχου πλευρά των κρατών μελών. Και εδώ είχε ένα ρόλο να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμως και τα ε, ηθικά κριτήρια, διότι ε, ποια από πού προέρχονται, πώς εξορίσονται οι πρώτες ύλες, ε, να δούμε ποιες κοινωνικές συνθήκες ε, επικρατούν. θα πρέπει να προσθέσουμε αυτό το κώδικα δεντολής, αυτά τα κριτήρια αν θέλετε, για την επιλογή των πρώτων ύλων. Λοιπόν, στην Ήτρε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων και κυρίως για την ετικετοθεσία και τα σχετικά κριτήρια. Ευχαριστούμε. Σαντούζα Τσίλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την σημερινή συζήτηση. Ε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Επιτροπή σα για την ε, μακροχρόνια υποστήριξή σα για αυτή την οδηγία, όπως τόνισαν πολλοί, οδήγησε σε μεγάλη εξοικονόμηση πόρων ναι, μια σειρά ετών. Ε, θα ήθελα να, ε, απηχώντας διάφορα σχόλια, να σχολιάσω πρώτα απ' όλα την ε, που σημαίνει σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων, όντω 45 ε, χρόνια χρειάζεται για να εφαρμοστεί σωστά ένα μέτρο. Απαγορεύονται προϊόντα πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κάτι δύσκολο. Ε, ε κάνουμε αξιολόγηση αντικτύπου, ε, αποτιμούμε τα μέτρα, χρειάζεται χρόνο, είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Όντω, σε ορισμένε περιπτώσει μπορούμε να επιταχύνουμε. Για την αυτή ε, μπορούμε όντως να συμπεριλάβουμε περισσότερα μέτρα ε, για τα ψυγεία, για τα πλυντήρια πιάτων, ε, για τα πλυντήρια ρούχων. Ε, προτείνουμε μέτρα και προδιαγραφές ε, για να παρατείνουμε το, το σχέδιο, το κύκλο ζωής ε, του προϊόντος. Οι εγγυήσει ε, που συνοδεύουν την αγορά ενός προϊόντος είναι ένα μέτρο που μπορούμε να υιοθετήσουμε για τις ηλεκτρικές σκούπες ή για τους λαμπτήρες, παραδείγματος χαρή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερα ε, δύσκολες δοκιμές ε, και συνεπάγεται και μεγάλο κόστος, οπότε μπορούμε να μελετήσουμε αυτή την ιδέα, αλλά ε, θα πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε την εφαρμογή των μέτρων σε σχέση με το προϊόν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση από πλευρά των εταιριών. Και αυτό με φέρνει και στο θέμα της ε, εποπτείας. Ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα, τις δραστηριότητες ε, και παρακολούθησης κοινής εποπτείας. Πριν από τα Χριστούγεννα κατατέθηκαν οι προτάσεις για το πακέτο για την παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που τώρα ακολουθεί τη συνήθι νομοθετική διαδικασία και τα πορίσματα αυτής της διαδικασίας θα επηρεάσουν και την οδηγία του οικολογικού σχεδιασμού. Α, τα κινητά. Ε, είπαμε στο σχέδιο δράσης, επειδή το αναφέρατε και στις πολλές φορές, πως ε, ε, θα πρέπει να λεπτομερέστερα να ασχοληθούμε με τα γεννητά γιατί αυτά τα προϊόντα σε σχέση με άλλα προϊόντα πληροφορικής αλλάζουν ραγδαία και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ώστε να ε, χειριζόμαστε αυτά τα προϊόντα που γνωρίζουν αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Η οδηγία για την ενεργειακή τοκητοθεσία που εγκρίθηκε πέρσι ε, Λοιπόν, το Κοινοβούλιο επέμεινε ιδιαίτερος ε, να μην επιδεινώνεται η απόδοση του προϊόντος ε, με τις αναβαθμίσεις του λογισμικού. Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να επιδιώξουμε και τώρα. Παράταση του κύκλου ζωής ήδη σήμερα... Βλέπουμε ε, μέτρα για τα ντους, παραδείγματο χάρη, για ό,τι σχετίζεται με κατανάλωση νερού ε, ή γενικότερα με ε, κατανάλωση ενεργειακών πηγών. Αλλά για τα προϊόντα που δεν τα μη ενεργειακά προϊόντα θα πρέπει να έχουμε προδιαγραφές ε, κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους. Αυτό είναι πολύ δυσκολότερο να το παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω στους εμπειρογνώμονες γιατί ε, υπέβαλαν ερωτήματα με τα μέλη της Επιτροπής ε, η κυρία Γκροστέτη, η κυρία Ριβαζή. Θέλετε να απαντήσετε. Η κυρία Ντράμπικ. θετική συζήτηση προκύπτει ότι θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε προδιαγραφές για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα που να είναι εφαρμόσιμες, όμως χρειάζονται περισσότεροι πόροι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στις Εθνικές Αρχές Εποπτείας, διότι ε, οι απαιτήσει ε, για την παρακολούθηση και η επέκταση του πεδίου αυτό συνεπάγονται αύξηση του κόστους Αυτό επίσης μπορεί να ε, δημιουργήσει και θέματα ανταγωνισμού εάν ε, για προϊόντα που προέρχονται ε, από τρίτες χώρες. Για την ανακύκλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επικρατήσει ε, στην αγορά, δηλαδή να εισάγει πρώτες ύλες ε, και να μεταποιεί στη συνέχεια τα προϊόντα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η εξαγωγή ε, αυτών των προϊόντων στη συνέχεια μπορεί να έχει κοινωνικές επιπτώσεις τρίτες χώρες. Sí, hay diversos aspectos que se han comentado. Uno que había incidido anteriormente Κοιτάξτε, πολλά υπόθηκαν. Εγώ θα ήθελα να πω πράγματα τα οποία σχετίζονται με αυτά που μελετήσαμε εμεί. Δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή αγορά εισάγει και προϊόντα και πρώτες ύλε. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα περισσότερο από ποτέ να λάβουμε υπόψη μας το θέμα των υλικών, γιατί εισάγουμε τα υλικά αυτά από τρίτες χώρες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις οι δικές τους ενεργειακές πολιτικές και οι πολιτικές μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος δεν ακολουθούν την ίδια διαγραμμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να τα πω πιο καθαρά και ξεκάθαρα ακόμα τη στιγμή που εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε ένα ποσοστό, ας πούμε να εφαρμόσουμε ένα ποσοστό ανανεώσιμων πηγών, έτσι όπως ε, προτείνει η ευρωπαϊκή πολιτική τη στιγμή που στη φάση της χρήσης εμείς είμαστε σε θέση ε, βάσει και των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουμε την ε, κατανάλωση παραδοσιακής ενέργειας έχουμε ενέργεια από κρίσμα μέταλλα σε πολλές περιπτώσεις τη στιγμή της δημιουργίας τους και της επεξεργασίας τους σε τρίτες χώρες χώρες οι οποίες βασίζουν το ενεργειακό τους μίξ σε το μείγμα σε ορυκτά ε, ε, ε, υλικά και σε παράγουν ενέργεια λοιπόν από ορυκτά θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό. Θα πρέπει να το, θα πρέπει να το μελετήσουμε. Και τα παραδείγματα είναι πολλά και εύκολα. Ε, ας πούμε, μπορεί κανείς να αγοράσει χαλκό, ας πούμε, από τη χιλή. Στη δεκαετία του 90 ο Χαλκός στην, ε, ε, ε, στην Χιλή ήταν στην επιφάνεια σε ποσοστό 3%. Τώρα αυτό έχει μειωθεί στο 1% και επομένω έχει εντετοκοποιηθεί η διαδικασία εξόριξης και αυτό, αυτή γίνεται με ένα ηλεκτρικό μείγμα ε, και χρήση ε, φυσικού αερίου. Επομένως ε, μιλάμε για χρήση ορυκτών πρώτων Εν πάση περιπτώσει έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε ότι η ανάλυση θα πρέπει να ε, ε, αφορά πλέον όλες τις διαδικασίες και όλες τις στιγμές ε, του κύκλου ζωής. Όσον αφορά την επισκευή των προϊόντων, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επισκευής, θα πρέπει να επεκταθεί ε, η ζωή των προϊόντων. Ε, υπάρχουν ε, πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει όχι από εμά, αλλά από άλλους πριν από εμά, όπου συγκρίνονται τα πλεονεκτήματα της επιμήκυνσης του, της ζωής ή ε, η επιλογή άλλων προϊόντων που μπορεί ενεργειακά να είναι πιο αποτελεσματικά. Ε, γίνονται στη μελέτη αυτή την οποία έχω κατά νου ε, κάποιες σκέψεις και ε, ε, καταλήγουν στο ότι 5 και 10% μπορεί να κερδίσει κανείς μέσω της επέκτασης του κύκλου ζωής. Ε, όχι μονάχα για τα νέα προϊόντα, αλλά και σε προϊόντα τα οποία μπορούν να υπάρχουν ήδη και για τα οποία απλώς θα επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής. Όπως ακούστηκε και από κάποιες, ε, ε, σε κάποιες παρεμβάσεις είναι πολύ σημαντικό και το προσυπογράφουμε η δυνατότητα ύπαρξης ανταλλακτικών να προωθήσουμε δηλαδή προϊόντα και αγορές ε, για τα οποία θα υπάρχουν ανταλλακτικά. και το σημαντικό στην ε, οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ε, ε, σημαντικό είναι να προβλεφθούν μέτρα για την αποσύνθεση των προϊόντων. Να είναι δυνατή δηλαδή αυτή η αποσύνθεση. Αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι υπάρχει και προγραμματισμένο τέλος ζωής για, το, για την καινοτομία ε, δηλαδή που μερικά ε, γίνονται πεπαλαιωμένα πριν φτάσουν και στην αγορά. Και ο, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο από άποψη περιβαλλοντική είναι υπογραμμίζοντας την δυνατότητα αποσύνθεσής τους και επομένως επαναχρησιμοποίησης των ανταλλακτικών τους. Εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, αυτά τα ανταλλακτικά τα οποία υπάρχουν στα προϊόντα αυτά, τότε δεν θα έχουμε χάσει τα υλικά λόγω ακριβώς αυτής της, προ... αυτής της πρώιμης ε, ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής που είναι κάτι διαφορετικό από, από το προγραμματισμένο τέλος του κύκλου ζωής. Εγώ επιμένω λοιπόν στο θέμα της δυνατότητας επισκευής, της δυνατότητας ε, επανάχρησης ε, της ε, συσκευής μέσα από κάποιες διορθώσεις ή κάποιες ανατάξεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ρής, λοιπόν, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Παρακαλώ, κυρία Ρής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη στη, στη συμπερισματική μου ε, τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την συζήτηση και έδωσαν ε, τα πολύτιμα σχόλιά τους. Ε, ο, ο βαθμός φιλοδοξία είναι πάρα πολύ ψηλός, ο βαθμός συνεκτικότητας επίσης πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θέλουμε ε, όλοι να συμμεριστούν αυτήν την φιλοδοξία και οι χρήστες και οι κατασκευαστές. Επίσης έγινε λόγος για τη στρατηγική αντιμετώπιση του κύκλου ζωής όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής και ανακύκλωσης. Ε, τα ερωτήματα της κυρίας Γκροστέτα βρίσκονται ήδη στην ε, ε, έκθεση το θέμα της επισκευής, επισκευασιμότητας, ας την πούμε έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ανέφερε και στην απάντησή του ο εμπειρογνώμονας πριν από λίγο. Όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ήδη το προτείνω. Γιατί λέω ότι δεν πρέπει να δούμε μονάχα την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ε, η κυρία Νταλίτα είπε νομίζω αυτά, ε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να δούμε ε, την δυνατότητα ε, χρήσης αλλά ε, να μην πολυβαρύνουμε το πράγμα το είπε και η κυρία Ούκενα δηλαδή να μην βάλουμε ένα σωρό ε, ένα σωρό προϋποθέσεις που δεν θα μπορέσει η αγορά να τις, να τις σηκώσει κατά κάποιο τρόπο, δεν θα μπορέσει η αγορά να ανταποκριθεί. Υπάρχουν ήδη μια σειρά προτύπων και στοιχείων προσημόρφωση. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να πούμε τι πρέπει να κάνουμε βράχη πρόθεσμα, τι μπορούμε να κάνουμε μάκρο ή μέσο πρόθεσμα. Θα πρέπει να δούμε λίγο αυτή τη χρονική γραμμή και τη χρονική αντιστοίχηση. Χρειάζεται λοιπόν φιλοδοξία, το είπαν και προηγούμενοι ομιλητέ. Εμεί την έχουμε την φιλοδοξία αυτή. Ο κύριο Κατάινεν ήταν όντω παρόν είναι γεγονός ότι όμως δεν συμμερίζονται όλοι ακριβώς την ίδια άποψη και τον, την ίδια ζέση. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε προς όλες τις καθε... κατευθύνσεις. Ευχαριστώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 6 Μαρτίου στις 11. Ψηφίζουμε στις 25-26 Απριλίου στην Επιτροπή. Επόμενο θέμα μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του προγράμματος live. Έχουμε διάφορους συνεισηγητές. Θα τους δώσω το λόγο. Αν είναι παρόντες βέβαια. Okay. So, I start with the, the co-rapporteurs or, the, or people representing them. So... Λοιπόν, ο κ. Καμπούς για την κυρία Σοβίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη, δεν, μπορούσα να δεν μπορεί να είναι η συγκεκριά παρούσα. Και θα μιλήσω όμως εξ ονόματός της. Έλεγε ότι ως σύμπροεδρος της ομάδας εργασίας LIFE, ε, η οποία από την αρχή της θητείας ασχολήθηκε με το θέμα, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συνεισηγητές για την ε, συμβολή του. Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό εργαλείο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ε, το ε, κλίμα και το περιβάλλον και που έχει στόχο ε, την υλοποίηση, βελτίωση κλπ. της ευνοσιακής πολιτικής όσον αφορά το κλίμα μέσα από συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που παρουσιάζουν προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ενδιάμεση λοιπόν ε, ε, επισκόπηση με αξιολόγηση των δύο πρώτων ετών του LIFE 14-16 και με αντίστοιχες προτάσεις σχετικά με την βελτίωση της κατάστασης. Σύμφωνα με την κυρία Σουίκα. Σουίτσα δίνονται πολλές πληροφορίες λεπτομερείς και απαραίτητες για την ε, μελέτη της, ε, της κατάστασης. Επίσης, ε, ζητούμε περισσότερες, περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματική χρήση όλων των πόρων, έτσι ώστε να υπάρχουν επομένως όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσει να γίνει η ενδιάμεση αξιολόγηση σωστά. Θέλει επίσης να υπογραμμίσει ότι δύο χώρες μέλη μοιράζονται παραπάνω από το 2 τρίτα του προπολογισμού LIFE για, το, για την περίοδο 14-16, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωστή κατανομή, η κατανομή των πόρων μεταξύ των χρόνων. Το LIFE είναι ε, σημαντικό εργαλείο για το κλίμα και το περιβάλλον και η κυρία Σουίκα ε, συμπρόεδρο τη ομάδα εργασία ε, για το LIFE θέλει και ευελπιστεί ότι θα βελτιωθούν και τα προγράμματα καθώς επίσης και οι διαδικασίες πληροφόρησης Επίσης ε, η κυρία Σουίκα μου έλεγε ότι ε, θα ήθελε να ζητήσει από τα, μέτρα, από τα μέλη της Επιτροπής ε, ε, Περιβάλλοντος να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας LIFE γιατί είναι απολύτως πεπισμένοι ότι το πρόγραμμα LIFE μπορεί να είναι εξαιρετικά καλό για τις χώρες μέλη και θα πρέπει ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να το υποστηρίξουμε το πρόγραμμα LIFE. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα ήθελα απλώς για μια ακόμα φορά να σας συγγνώμη εξ με τη κυρία Σουίκα η οποία δεν μπόρεσε δυστυχώς να είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πότσεκ, μέρος του κύριου Καπούτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφο μου Νίκολα Καπούτο δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα. Μου ζήτησε να εκφράσω κάποια σχόλια γνωστού. Αυτό είναι μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, δεν διαβεβαιώσει. Το πρόγραμμα LIFE. ακολουθεί σωστό δρόμο, θα είναι αποτελεσματικό, διότι έχει καλού στόχου ε, και στόχου κλιματολογικού περιβαλλοντικού και βασίζεται στη στρατηγική τη Ευρώπη για το 2020. Μετά είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα, διότι τα προγράμματα θα, προθήσουν, θα δώσουν κάποια αξία για τι επενδύσει. Το όφελο για την κοινωνία κάποιων προγραμμάτων τον διαγωνισμό του 2014 αναλογούν σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το στοιχείο από μόνο του είναι τέσσερις φορές ε, το κόστος ε, του προγράμματο ε, live για το 2014 επειδή τα προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί αντιμετωπίζουν προβλήματα, δηλαδή η απώλεια η οικονομία από την κυκλική οικονομία, μείωση του κόστου έλλειψης δράσης όσον αφορά ε, την αλλαγή του κλίματος και μετά έχουν συμπληρωματικά αποτελέσματα διότι ε, συντονίζεται με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης το LIFE όμως η εξολόγηση επίσης ε, τονίζει και πτυχές οι οποίες χρήζουν βελτιώσεων δηλαδή πρώτα απ' όλα απλούστευση διαδικασιών ελέγχου χορηγιών, υποβολή αιτήσεων, υποβολή εκθέσεων, πιο δίκαιη κατανομή και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πόρων του LIFE μεταξύ κρατών μελών. Δύο κράτη-μέλη έχουν πάνω από το 1 τρίτο των πόρων του LIFE για την περίοδο 2014-2015. Πρέπει να ισχυθεί ο ρόλος των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, των ενώσεων για να προτίσουν, για να υπογράψουν και να δρομολογούν τα προγράμματα αυτά. Χρειάζεται βελτίωση της ε, στατικής επικοινωνίας για καλύτερη στόχευση του ακροτηρίου και θα πρέπει να στέλνουμε μηνύματα με βάση τους στόχους και τα αποτελέσματα χρειάζεται διαθρωμένος συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Και κυρία Πρόεδρε, αν με επιτρέπει Πρόεδρος, πέραν αυτών που λέει ο συνάδελφος ο κ. Νίκολα Καπούτο, θέλω και εγώ να προσθέσω κάτι όσον αφορά την αξιολόγηση ότι πρέπει να δούμε και το πρόβλημα του όγκου της χρηματοδοτήσεως. Οι πόροι του LIFE αντιπροσωπεύουν μόνο 1,03 του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσης, άρα είναι ανέφικτο να πετύχουμε όλες τις, τους στόχους, τους μακροπρόθεσμους. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ, εκ μέρους της. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Μάργαρετ υποστηρίζει το περιεχόμενο του ψηφίσματος που εξετάζεται από την Επιτροπή και τα συνοδευτικά ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνεται υπόψη, αρκετά υπόψη, σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξολόγηση. Έχουμε ανησυχία όσον αφορά την έλλειψη στατιστικών αναλυτικών στοιχείων για να γίνει σωστή αξιολόγηση του ΛΑΙΦ. Λείπουν οι λεπτομέρειε και πιστεύουμε ότι το ψήφισμα και η προφορική ερώτηση διερευνούν αυτά τα βασικά στοιχεία. Καταρχάς, δίνεται προτεραιότητα στην κατανομή των πόρων όχι μόνο για τα αυτονόητη απέτηση για δίκαιη κατανομή αλλά χρειάζεται ένα πιο δίκαιο σύστημα και αποτελεσματικότερα αποτελέσματα. Δεύτερον, δίνεται σημασία σε πλέον ολοκληρωμένη και συμβιωτική προσέγγιση για τα προγράμματα έτσι θα μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα και θα μαδοποιούνται οι πόροι και αυτό καταλητικά θα επηρεάσει την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων θα κινούνται σε ανώτερο επίπεδο, όχι μόνο τοπικό. Ε, υπάρχει έλλειψη στοιχείων για να αξιολογηθεί η επιτυχία και τα κενά του προγράμματος. Χρειάζονται αυτά τα στοιχεία, ε, ώστε στον επόμενο γύρο του προπολογισμού να μπορούμε να δικαιολογήσουμε μια συνέχιση του προγράμματος LIFE ή κάτι, κάποιο αντίστοιχο προγράμματος. Και για το σχεδιασμό μετά το LIFE Θέλουμε να γίνει σωστή ανάλυση των προγραμμάτων που ήταν αποτελεσματικά και θα πρέπει να επαναληφθούν οι βέλτιστες πρακτικές, οι εξοικονομήσεις και η στήριξη κατά πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Εκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πάντοτε προσπαθούμε να προσφέρουμε αμοιβαία υποστήριξη, να καταλήγουμε σε συμφωνίες, ούτως ώστε να βελτιστοποιούμε τα αποτελέσματα στις εργασίες μας. Επίσης, το πρόγραμμα ε, LIFE συνδέεται με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τη γεωργία ή την ε, πολιτική συνοχής. Όταν προετοιμάζαμε ε, την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ψήφισμά μας, είχα διευκρινίσει ότι σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε σε αυτές τις δύο πολιτικές. Χωρίς όμως ε, καταλήξη αιτιολόγηση, συγγνώμη, απερίφθη αυτή η πρόταση από τους ε, συνεισηγητές. Ε, βλέπουμε ότι με την πολιτική γεωργίας, ε, κυρίως τους συντηρητικούς συναδέλφους, πολύ ε, σπασμωδικές αντιδράσεις. Υπάρχουν ε, πολλοί άριθμα προγράμματα που χρηματοδοτούνται ε, και που συνδυάζουν ε, την προστασία του περιβάλλοντος και τη γεωργία. Με αγνόησαν όμως. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει αυτές τις συνέργειες άμεσα στο LIFE και σε άλλα προγράμματα ε, διότι αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό της καλλιεργούμενης γης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλαβαίνουμε πόσο κέριος είναι ο ρόλος των δράσεών μας για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Λοιπόν, ε, όταν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE μπορούμε να βρούμε τρόπους να προστατεύουμε και το περιβάλλον, η κατάσταση είναι win-win και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε αυτή την στάση να τηρήσει. Σας ευχαριστούμε κάποιο άλλος. Όχι, ο κύριο Δεγάντο Ρώσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή ΕΜΒΗ ε, για αυτό τον πολύ επικοδομητικό διάλογο για το πρόγραμμα LIFE. Το LIFE άρχισε το 92, έχει 25 χρόνια ζωής ήδη και εν γέννη θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα πέντε ε, κύκλους έχει περάσει ε, και με το feedback, με τις αξιολογήσεις ε, που γίνονται, το αναβαθμίζουμε διαρκώς. Για την περίοδο 2014 και 2020 στην ενδιάμεση αξιολόγηση είδαμε λοιπόν που ήταν θετικά τα αποτελέσματα. τα προγράμματα LIFE είναι πολυετή και Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία το 2000, περιμένουμε περισσότερα στοιχεία το 2016 όταν κάνουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση και πολλά προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με το LIFE, απλώς ε, τα προγράμματα έχουν το δικό τους ρυθμό και αυτό δεν μας εμποδίζει το να προσδιορίσουμε ποιο είναι το ετήσιο κόστος και ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ε, θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα κάθε πρόγραμμα. Πάντως, στην ενδιάμεση αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε ότι αυτά τα προγράμματα Life Integrated, που είναι μια δοκιμή, ένα νέο στοιχείο που δοκιμάσαμε, ε, όπου προσφέρεται αερογή προς τα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν βασικές με βασικά περιβαλλοντικά νομοθετήματα και εδώ παραθετικά να πω πως ε, υπάρχουν αυτά τα προγράμματα στόχοι που καλύπτουν το, το, ε, την ποιότητα του αέρα, την ε, προσαρμογή για το περιβάλλον, την προστασία της γης σε μεγάλες ευρύτατες γεωγραφικές περιοχές, πολλές πόλεις, περιφέρειες, περιοχές και πρόκειται για δράσεις που υπερβαίνουν το πεδίο του προγράμματος. Αυτό ε, συνεπάγεται η κινητοποίηση αξιωμένης χρηματοδότηση που προέρχεται κυρίως από άλλα ε, ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεπάγεται και περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή, αυτό είναι το νόημα της ε, συνέργειας και του καταλητικού ρόλου που έχει το LIFE. Επίσης, στην ενδιάμεση αξιολόγηση εντοπίστηκαν δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτό το πρόγραμμα, απλούσταση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων. Αυτό συνέβη ήδη ε, για αυτή την τρέχουσα περίοδο μέχρι το 2020 μέτρα επίσης που τονίζουν το καταλητικό ρόλο των προγραμμάτων και Υπάρχουν και διάφορα ζητήματα που θα συμπεριληφθούν ε, στην πρότασή μας για τη συνέχιση του LIFE μετά το 2020. Θα συνοδεύονται από μηχανισμούς για τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κυκλική οικονομία Φερρυπίν. Θα χρειαστεί χρηματοδότηση μια κρίσιμη μάζα ε, και γίνεται αξιολόγηση τώρα αντικτύπου για το την περίοδο μετά το 2020 για να καλύψουμε και αυτό το θέμα που αναφέρατε κι εσείς ε, για την ε, ομοιόμορφη απορρόφηση των κονδυλίων του LIFE ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, ούτε και το προηγούμενο σύστημα των εθνικών κονδυλίων, ούτε και το νέο σύστημα των σωματωμένων προγραμμάτων επέτυχαν τον στόχο αυτό της ομοιόμορφης απορρόφησης κονδυλίων. Λοιπόν, προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ώστε να μετεξελίσσεται ε, διαρκώς το ΛΑΦ για να καλύψει ε, τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και κλείνοντας να σας πω ότι δεδομένου του περιορισμένου προϋπολογισμού του LIFE μπορούμε να περιμένουμε να καλύψει όλες τις ανάγκες μας για το κλίμα και για το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να επιδιώκουμε ενσωμάτωση αυτών των προγραμμάτων σε πολιτικές. Ε, γίνονται οι παρεμβάσεις μέσω του ΛΕΦ για να καταδεικνύονται ποιες είναι οι προσφορότερες λύσεις και για να λειτουργεί καταλητικά για αυτά τα ενσωματωμένα, τα ολοκληρωμένα προγράμματα στα οποία προαναφέρθηκα. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ε, θέλει κάποιος ε, να επανέλθει. Όχι. Καταληκτική ημερομηνία για τις, προθ... για τις τροπολογίες 6 Μαρτίου ε, στις 11 και 26 ε, και 27 Μαρτίου στην ΕΜΒΗ θα ψηφίσουμε. Πάμε στο τελευταίο σημείο της μερικής διάταξης. Ε, εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης της Μαριάννα Πέτυρ για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νοσιακού δικαίου το 2016. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν η Κροατία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότεροι πολίτες που ήθελαν να μπει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσαν το κράτος δικαίου ήταν ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από όταν έγινε μέλος η Κροατία το κράτος δικαίου πάντα ήταν ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα και από όταν γίναμε ανεξάρτητοι. Μπόρεσα να αξιολογήσω ότι αυτό ίσχυε και για ε, κατοίκους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Διότι ο σεβασμός των νόμων είναι σημαντικότατο στοιχείο. Αν εφ' αυτού δεν υπάρχει ασφάλεια, επενδύσεις, πρόοδος, δεν υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Βάσει αυτών ήθελα να πω ότι ήταν σημαντικό η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Έτσι προστατεύονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσης και δημιουργείται και πολύ θετικό κλίμα για τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι κάτι απαραίτητο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας το 2016 αναφέρεται σε αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων και αναφέρεται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν θα τονίσω το εξής. Η αύξηση παραβιάσεων των δικαιωμάτων και του δικαίου το 2016 σε θέματα υγείας και παραβάσεις σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων αυξήθηκαν από το 2010 αυξήθηκαν το 2016 σε σχέση με το 2015. Πέραν αυτού είχαμε παραβάσεις σε διασυνοριακά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για θέματα περιβάλλοντος είναι περιπλοκότατη καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται σωστά κυρίως για την χρήση των προενταξιακών πόρων. Αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, η κατάσταση είναι καλή, αλλά χρειαζόμαστε αύξηση της διαφάνειας. Η παρούσα κατάσταση οδηγεί σε διαμαρτυρίες καταγγελίες. Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι καταγγελίες των Ευρωπαίων πολιτών για θέματα εφαρμογή εφαρμογής των ε, ευρωπαϊκών νόμων. Αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρονται περισσότερο οι πολίτες. Ε, οπότε η αύξηση των καταγγελιών δεν είναι κάτι κακό. Ε, σε θέματα υγείας, σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων υπάρχουν καταγγελίες δεν έχω αναφερθεί λεπτομερώς σε αυτά τα θέματα στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Θα καλύψω τα θέματα αυτά στις τροπολογίες και θα συνεργαστούμε πάνω σε αυτό με τους ε, σκιώδεις ηγητές. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις ηγητές, ο κ. Βόλκαν ο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφε, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Δυστυχώς, όμως, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι επειδή υπάρχουν ελλείψεις και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νοσιακού δικαίου, αυτό συνεπάγεται μεγάλο κόστος, ε, όχι μόνο πλευράς χρημάτων, λοιπόν, αλλά και ανθρώπινες ζωές, γιατί βέβαια, πεθαίνουν οι άνθρωποι για ε, χιλιάδες άνθρωποι λόγω της κακής ε, ποιότητας ε, του ατμοσφαιρικού αέρα επειδή ε, δεν εφαρμόζονται σωστά οι κατευθυντήριες γραμμές. Ε, είναι λοιπόν σοβαρότατο το πρόβλημα και θα πρέπει να διαπιστώσουμε επίσης ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός διαδικασίων επί παραβάση και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη και λένε κάποια κράτη-μέλη ότι «Α, σε μας δεν είναι τόσο κακή η κατάσταση», αλλά δυστυχώς εμείς διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα, κυρίως ε, στους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. 2016 υπήρχαν 1.671 διαδικασίες επιπαραβάσεις, 300 400 περισσότερες σε σχέση με ε, πέρυσι. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απαιτείται δράση. Ε, για τα κράτη-μέλη... Ε, απαιτείται ε, αμελητή να εφαρμόζουν σωστά ε, το ενωσιακό δίκαιο. Γιατί αυτές οι κατευθυντήριες γραμμέ για την ποιότητα του αέρα ήταν από το 2010 παραδείγματο χάρη. Χρειάζονται υπερβολικά πολύ χρόνο για να μεταφέρουν την οδηγία. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το επιχείρημα ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Επίσης, ε, για την παρακολούθηση των οχημάτων, αν υπήρχε ε, μεγαλύτερη νοσιακή αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα, σίγουρα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα για την ε, προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Βλέπουμε ότι δεν ε, επαρκεί λοιπόν η διαδικασία επί παραβάση. Δηλαδή εμείς πολύ ολαιότατα νομοθετήματα να φτιάχνουμε εδώ πέρα, ε, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κιόλα. Δηλαδή πέρα από τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες μας ε, θα πρέπει να ασχολούμαστε επισταμένα με την εφαρμογή τους. Και θα ήθελα απευθυνόμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι χρειάζονται υποστήριξη τα κράτη-μέλη ορισμένες φορές και στα κράτη-μέλη θα ήθελα να πω ότι μιλάμε για, συζητούμε για τον νέο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, οπότε θα πρέπει να προβληματιστούν τα κράτη-μέλη μήπως ε, στην τοποθέτησή τους για τον νέο προπολογισμό και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ε, δεν θα έπρεπε να ε, αναδείξουν σε προτεραιότητα και πάλι την προστασία του περιβάλλοντος Χρειαζόμαστε ε, συλλογικούς ε, τρόπους ε, παρακολούθησης εφαρμογής των νομοθετημάτων γιατί αυτό χρειάζονται οι πολίτες και νομίζω ότι αυτό θα υποστήριζε και τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Άλλος, ο κ. Κέρκ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Α, είναι. Έχετε το λόγο. Ο κ. Σλούτσιος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μέλη του Κοινοβουλίου. Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις της Επιτροπής. Συνάδουν αυτά με αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Ευπρόσδεκτη γενική υποστήριξη για τη νέα πολιτική να κινούμεθα ταχύτερα όσον αφορά τις περιπτώσεις παράβασης. Το περιβάλλον είναι τομέας προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. διαβεβαιώνω. Ευχαριστώ. Η κυρία Θέλετε να προβείτε σε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα τα στοιχεία αυτά που ανέφερα στην εισαγωγή μου απαιτούν μία κάποια αντίδραση και πιο στενή στην εργασία με τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν είμαι υπέρ της επιβολής κυρώσεων. Τα πιλωτικά προγράμματα είναι πολύ καλά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όλα τα κράτη-μέλη καλούνται, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις οδηγίες και να τις ενσωματώσουν στη δική τους ένωμη Όσον αφορά το περιβάλλον υπάρχουν πολλά προβλήματα και μπορούμε να σημειώσουμε ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους ότι μπορούν να συμμετάσχουν, μπορούν να προσφύγουν σε περίπτωση παραβάσεων. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν. Κοινοβουλευτικές επιτροπές, το Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, οι πολίτε και οι επιχειρήσει πρέπει να συνεργαστούν και έτσι μπορούμε να πετύχουμε με αυτή τη συνεργασία τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Το περιβάλλον το οποίο θέλουμε να το αφήσουμε σε καλή κατάσταση και για τι μελλοντικέ γενιέ. Ευχαριστώ. Ακριβώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πετήρ. Εδώ ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας, τα απογεύματος. Θα τα πούμε σε 9. Για την γνωμοδότηση της κυρίας Πετήρ, προθεσμία. Είναι 1η Μαρτίου στις 11 για τροπολογίες και στις 27 Μαρτίου ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.